So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte doch die Plätze einzunehmen. Wir haben ja ein bisschen. Έχει αλλάξει λίγο το χρονοδιάγραμμα σήμερα. Αρχίζουμε παρατέταρτο και ευθύ αμέσω με την ψηφοφορία. Μετά έκθεση Wilmot, αμέσως μετά την ψήφο. 17 και 30, 18 και 30 θα είναι παρόν εδώ ο Επίτροπος κύριος Ταγιάννη και από 18 και 30 έως 19 και 15 έκθεση Μπαρτολούτσι για τους συσσωρευτές. Ας αρχίσουμε λοιπόν αμέσως. Τοποθετήστε τις ε, κάρτες ψηφοφορίας ή ζητήστε να σας τις φέρουν, εάν ορισμένοι δεν τις έχετε. Και αρχίζουμε με την έκθεση Παναγιώτο. Πρώτη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών δύο ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Παρακαλώ ψήφι υπέρ αντίθετη, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9, ο εισηγητής είναι υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Block vote, τροπολογίες 12, 14, 15, 16, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 3 υπέρ. Συμβαστική δηλαδή. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφιστεί 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Θα ψηφίσουμε ονομαστικά, δηλαδή ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία 17. Ψηφίσατε παρακαλώ. Πέρας. 16 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ας ψηφιστεί ονομαστικά και η 13 λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται με 30 ψήφους υπέρ και 15 κατά. ...47 και 48... ...ορίστε αλλά δεν έχει μικρόφωνο... ...η παρεμβαίνουσα. Βάλτε καλά την κάρτα σας μέσα... ...αλλιώς να αλλάξετε θέση. Αν δεν... ...πετυχαίνει αλλάξτε θέση παρακαλώ. Και στο μεταξύ θα κοιτάξουμε να διορθώσουμε το μηχάνημα. Block vote λοιπόν 47-48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, εγκρίνονται μάλλον. Τροπολογία 4. Με συγχωρείτε. 5. 5. Φύγα κάπως πολύ γρήγορα. Ψήφι υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ας ψηφιστεί λοιπόν ηλεκτρονικά ψηφίσατε πέρασε. σαφώς θετικό το αποτέλεσμα. Τελική ψηφοφορία. Κύριε Γκροστέτ. Δεν λειτουργεί Έρχεται ο τεχνικός, κυρία συνάδελφε, ναι. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Αυτή τη στιγμή λέει ο πρόεδρος. Να επαναλάβουμε την τελευταία ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν πάλι την τροπολογία υπαριθμών 24, όπως είπα η ηλεκτρονική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται η ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία. ηλεκτρονική όπως είπα, αρχίζει, ψηφίσατε, τέλος. 51 ψηφί, υπέρ, καμία κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν, συγχαρητήρια κύριε Σιγητά, δεν τελείωσε όμως η ώρα των ψηφοφοριών έχουμε, ούτε καν η ψηφοφορία αυτή, έχουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Στο σύνολό του, ηλεκτρονικά πάλι, αρχίζει η ψηφοφορία, ψηφίσατε παρακαλώ. Πέρα. Εγκρίνεται. Επίσης, θα δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή, διότι έχουμε το νέο άρθρο 70. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μεγάλη επιτυχία για όλους, διότι το θέμα αυτό χρονολογείται το 2006, ίσως και πιο πριν. Ήταν λοιπόν ιδιαίτερα επίμαχο, αμφιλεγόμενο θέμα, είχε κολλήσει, δεν προχωρούσε. Ευτυχώς επιτέλους χάρη στους Σλούτερ, Κούκοβιτς, Γιόργενσεν, Ρόσκι, Μαστάρκε, Γκρίς βεβαίως και σε όλους τους άλλους που συνεργάστηκαν, συνεργάτες των βουλευτών κτλ. Απέβει μεγάλη επιτυχία για το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι συνδυάζει κοινωνικά, οικονομικά, τεχνολογικά και πολιτικά θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για την εργασία που επιτελέσατε εσείς, διότι βέβαια κάποιος πρέπει να κατευθύνει το σκάφος ως πλοίαρχος, ας πούμε. Ρωτώ τώρα λοιπόν, θέλετε να ζητήσετε ψηφοφορία εντολής, οπότε χρειάζεστε πλειοψηφία 35 ψήφων για να μπορέσετε να προχωρήσετε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Βλέπω ότι νεύεται καταφατικά. Θεωρώ λοιπόν ότι μου λέτε ναι και θα κάνουμε την ψηφοφορία αυτή. Επίσης ονομαστικός δηλαδή ηλεκτρονικός και αρχίζει η ψηφοφορία τώρα. Ψηφίσατε. Πέρας. Τι να ζητήσει κανεί καλύτερο. Το βλέπετε το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια λοιπόν. και Παναγιώτοφ, καλή επιτυχία στις διαπραγματεύσεις. Βεβαίως θα είμαι και εγώ κοντά σας και θα έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε τακτικότερα. Ερχόμαστε στην επόμενη ψηφοφορία, έκθεση Ρόσμπαχ. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 8 με ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εδώ θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει για το δεύτερο τμήμα ψηφίσατε πέρασε με μεγάλη πλουψηφία, υπέρ τροπολογία 9 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 32 εκπίπτει. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. 47. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. ...36 ψήφοι υπέρ 24 κατά... ...εγκρίνεται. Η κυρία Άουκεν. Δεν έχει μικρόφωνο η κυρία Άουκεν. Από ρεφλέξ αντιδρώ έτσι, λέει ο πρόεδρο. 48. Αν με συγχωρείτε. 47. Όχι, 48. 48 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. άποχέ, Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. άποχέ, Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 17. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος. 37 ψήφι υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. 18 υπέρ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 ε, γνωμοδοτήσεως της. Τώρα, πάλι η κυρία Ρόσπαχ για την περιφερειακή πολιτική και τις βιομηχανικές περιφέρειες της Ένωσης, τροπολογία 1, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται δύο υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. τρία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. τέσσερα υπέρ, αυτή η όχι ψηφίζεται. τέσσερα λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ας α, ε, επαληθευτεί λοιπόν. Ψηφίσατε. Πέρας. Σαφές το θετικό αποτέλεσμα. 5 υπέρ, κατά, άποχέ, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Α, συγγνώμη, απορρίπτεται, απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, άποχέ. απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε την 12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 Κατά. Φαίνεται να ψηφίζουν μόνο οι συνάδελφοι των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ψηφίζω λοιπόν ηλεκτρονικά. 23. Ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Πέρας. Σαφώς εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Βλέπετε το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια κύριε Ρόσπαχ. Ευχαριστώ για την αυτοπιθαρχία που δείξατε στην διάρκεια της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ όλοι να συμμετάσχετε στα clinical trials. Βεβαίως εφόσον υπάρξει κάποια ησυχία θα πάρει το λόγο η κυρία Wilmot. Έχουμε προβλέψει περίπου 45 λεπτά για την συζήτηση. Πρώτη λαμβάνει το λόγο η εισηγήτρια. Παρακαλώ, ωστόσο, κάντε λίγη ησυχία για να μπορέσει να μιλήσει η εισηγήτρια. Ich glaube, wir können jetzt starten. Glennis Wilmot hat jetzt ausschließlich das Wort. Bitte, Glennis, please. Glennis Wilmot hat das Wort. Ευχαριστώ Ματίας και ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους που έδειξαν ε, μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το νομοθέτημα. Η αναθεώρηση χρειάζεται έτσι ώστε να έχουμε ηγετική θέση στην έρευνα και θα πρέπει να μην έχουμε ε, καθυστερήσεις εξαιτίας της μεγάλης γραφειοκρατίας και να υπάρχει ασφάλεια και διαφάνεια. Είχαμε 700 τροπολογίες και θα ήθελα να σταθώ στα βασικά ζητήματα. Μερικές είναι πολύ καλές και υπάρχουν πιθανότητες και δυνατότητες συμβιβασμού. Ξέρω ότι πολλοί ασχολούνται με τις επιτροπές δεοντολογίας και αυτό είναι κάτι το οποίο με έχει απασχολεί. Γκρένης, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Μήπως θα είχατε την ευγενική καλοσύνη είτε να σταματήσετε να παρακολουθήσετε τη εισηγήτρια είτε να αποχωρήσετε. Όπως έλεγα, πολλοί ασχολούνται με τις επιτροπές δεοντολογίας, κάτι το οποίο με απασχόλησε. Νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια καλή θέση και στάση, αλλά θα πρέπει να φτάσουμε σε εξισορρόπηση χωρίς να είμαστε υπερδιεξοδικοί. Πολλοί υπέβαλαν τροπολογίες για μεγαλύτερη προθεσμία για τις κλινικές δοκιμές. Κατανοώ γιατί το έκαναν αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα χρονικά όρια της Κομισιόν. Ξέρω ότι είναι φιλόδοξα, αλλά βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ερευνητές μου ζήτησαν υποστήριξη. Επίσης, η μακροχρόνια διαδικασία μέχρι την έγκριση σημαίνει ότι χάνουμε μεγάλο τμήμα της αγοράς και περιμένουν και ασθενείς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν από τη θεραπεία. Γνωρίζω ότι ε, ζητήθηκε παράταση, γι' αυτό θα πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει καλή διαπραγματευτική θέση για να φτάσουμε σε καλό συμβασμό στο τέλος της συζήτησης. Ένα άλλο θέμα είναι οι χαμηλές κλινικές δοκιμές. Δηλαδή να χρησιμοποιούνται φάρμακα μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας εθνικής αδειοδότησης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει χρήση εκτός σήμανσης μέσα στα πλαίσια της χαμηλής παρέμβασης τη στιγμή που μιλάμε για ε, τυποποιημένες κλινικές πρακτικές. Δεν υπάρχει πολλές φορές άλλη δυνατότητα από την χρήση ε, φαρμάκων εκτός σήμανσης, διότι για ορισμένους ε, παιδικούς ε, καρκίνους δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ενώ για άλλους καρκίνους δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Για τους περισσότερους καρκίνους τα σκευάσματα είναι εκτός σήμανσης. Γι' αυτό θα ήθελα να είσαστε ανοιχτόμυαλοι επί του θέματος ως προς το σύστημα εθνικών αποζημιώσεων έχουν υποβληθεί ε, ορισμένες τροπολογίες και ξέρετε ότι ο κόστος ασφάλισης είναι πολύ, πολλές φορές αστρονομικό, ιδιαίτερα για σπάνιες ασθένειες. Γι' αυτό θα πρέπει τα χρήματα αυτά να πάνε στην έρευνα και όχι στα ασφάλιστρα. Και πολλές φορές η αποζημιώση είναι, η αίτηση αποζημιώσεων είναι πολύ ε, χαμηλού ύψους. Γι' αυτό υπάρχουν καλά ε, και αναγνωρισμένα σχέδια από τη Δανία και από άλλες χώρες. Ως προς τη διαφάνεια, αυτό θα το συζητήσουμε και με τους σκιώδεις, η ε, βιομηχανία πιστεύει ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και υπερβολική γραφειοκρατία. Θα Ήθελα να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει μεγαλύτερη διαφάνεια, διότι η έλλειψη διαφάνεια έχει μειώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα φάρμακα και οι επιστήμονες ε, μπορούν δύσκολα να φτάσουν σε αυτά τα συμπεράσματα και να ζητήσουν αναθεώρηση. Επίσης, πολλά ε, ερευνητικά, πολλές δοκιμές δεν έχουν δημοσιευθεί. Οι δοκιμές επαναλαμβάνονται πολλές φορές πριν δημοσιευτούν. Θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πέραν της πρότασης της Επιτροπής και να ζητήσουμε σύνοψη αποτελεσμάτων. Επειδή πολλές φορές υπάρχει μεροληψία, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ότι θα διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού για τα φάρμακα. Θα ήθελα να συνεργαστώ βεβαίως εκ του σύνεγγης και με τους σκιώδεις για όλα αυτά τα επιμέρους θέματα. Ευχαριστούμε Γκλένης. Εισερχόμεθα στην συζήτηση τώρα με τις κυρίες Παρβάνοβα, Άουκεν, Σάρμπενοχ και Αλτασούσα, που είναι οι σκιώδεις συζητητές. Πίτα Λίζε, Edith Estrada, Michel Ριβαζί, Kollegen Περιλό. Äh, Είναι τα ονόματα των υπολείπων εγγεγραμμένων. Η κυρία Ροσπά αναλαμβάνει όλα τα βάρη όλη τη πολιτική τη ομάδα. Α βάλουμε παντού Άννα Ροσπά. Μήπω μήπως δεν άκουσε κανεί το όνομά του που επιθυμεί να ομιλήσει. Ωραία. Τότε λοιπόν μπορώ να κλείσω τον κατάλογο των εγγεγραμμένων και θα δώσω από 4 λεπτά στους σκιώδεις συζητητές και μετά ίσως κατέβουμε στα 2 λεπτά. Γιούβεν. Ευχαριστώ πρόεδρε για αυτά τα 4 λεπτά. Το κείμενο είναι καλό και η εισήγηση ε, είναι πολύ καλή επίσης της ε, κυρίας Ούλμοντ. Τώρα, επί των συγκεκριμένων θεμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην ανακατέψει πολύ ε, την ε, ήδη υπάρχουσα αρχιτεκτονική δομή. Είναι πολύ καλή ιδέα και εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια προσέγγιση. Να μην φέρουμε τα πάνω κάτω στην οδηγία, να μην την αλλάξουμε ριζικά, μπορούμε βέβαια να τη βελτιώσουμε. Για παράδειγμα, για τις δοκιμές μικρής παρέμβασης. Δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Ε, εγώ μπορώ με μια τέτοια παρέμβαση να σκοτώσω κάποιον. Μια ένεση με δηλητήριο είναι υψηλού κινδύνου παρόλο που είναι χαμηλής παρέμβασης. Το θέμα είναι να είναι χαμηλού κινδύνου, όχι χαμηλή παρέμβασης. Μετά, οι επιτροπέ δεοντολογίας θα πρέπει να ξαναμπούν στο κείμενο. Το επιθυμεί το Κοινοβούλιο. Αλλά ας αντιληφθούμε ότι οι επιτροπές αυτές κάνουν πολύ διαφορετικά πράγματα από χώρα σε χώρα. Οπότε εμεί θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιο είναι το καθήκον του, ποια είναι η αποστολή του. Επίση, θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση για τι έκτακτε περιπτώσει. Ε, σε ό,τι αφορά το θέμα των ευάλωτων ατόμων, θα πρέπει να προστατευτούν ιδιαίτερα. Η δυσκολία είναι η εξή. Τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικό ορισμό για τα ευάλωτα άτομα. Θα πρέπει λοιπόν κατά κάποιο τρόπο να καταλήγουμε σε ένα περιορισμένο κατάλογο. Ένα σχόλιο μόνο σε ό,τι αφορά το τελευταίο σχόλιο της κυρίας Βίλμοντ, σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση δηλαδή. Καταρχήν, η διαφήμιση των δοκιμών να είναι υποχρεωτική. Ε, δηλαδή η, δημοσιοποίηση τους μάλλον να είναι υποχρεωτική. Γιατί ως τώρα δεν είναι υποχρεωτική. Καλό λοιπόν να γίνει υποχρεωτική. Δεύτερον, θα πρέπει να προσέξουμε τα λόμπι που θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα χωρίς να κάνουν τα ίδια τα λόμπι τις ε, δοκιμές. Συνεπώς, πρώτον, η δημοσίευση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, που δεν είναι σήμερα. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνεται με δύο τρόπους. Πρώτον, προς το κοινό, με έναν τρόπο δηλαδή κατανοητό, εύληπτο από το ευρύ κοινό, γιατί αν δώσουμε ε, πολύ λεπτομερή δεδομένα ενδεχομένω δεν θα τα καταλάβει καλά το κοινό, οπότε ε, μπορεί να μην πετύχουμε και το στόχο μας, να πετύχουμε τον αντίθετο ακριβώς. Συνεπώς μια συνοπτική δημοσιοποίηση καταρχήν για, το ευρύ κοινό και δεύτερον πληροφορίες θα είναι τα πορίσματα των ερευνητικών προσπαθειών. Εκεί αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι πολύ πιο πλήρεις. Ταυτόχρονα όμως προσοχή να μην δίνουμε όλα τα δεδομένα, το 100% διότι υπάρχουν κάποια λόμπι τα οποία έρχονται και μας ε, επισκέπτονται είναι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι δεν έχουν κάνει ποτέ μια κλινική δοκιμή οι ίδιοι, αλλά χρησιμοποιούν τι κλινικέ δοκιμέ άλλων. Δηλαδή κάνουν μετααναλύσει, αναλύσει στοιχείων τα, οποία αφορούν μελέτε που έχουν κάνει κάποιοι άλλοι. Δεν ε, θέλουμε να σπρώξουμε τους, τους πανεπιστημιακούς να μην κάνουν έρευνα, να μην κάνουν δοκιμές. Τέλος, Κάτι που φαίνεται λεπτομέρεια αλλά δεν είναι. Ε, η προθεσμία για τη δημοσίευση. Ε, η Κομισιόν λέει ένα χρόνο μετά το, το τέλος των δοκιμών. Ε, δυστυχώς αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται, όλοι το λένε, χρειάζεται τουλάχιστον δύο χρόνια για την πρώτη δημοσίευση. Οπότε θα πρέπει να το εξή, να δώσουμε δύο χρόνια για να δώσουμε ε, ε στους αναδόχους την ε, δυνατότητα να δημοσιεύσουν τα πρώτα αποτελέσματα σε ε, μια επιστημονική επιθεώρηση ε, που θα υπόκειται σε έλεγχο ομολόγων. Έτσι ώστε να συζητηθούν τα αποτελέσματα καταρχήν μεταξύ εμπειρογνωμόνων, μεταξύ ειδικών και δεύτερον οι πανεπιστημιακοί αφού θα έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους σε ένα επιστημονικό περιοδικό, δεν θα φοβούνται ότι κάποιος θα τους τα κλέψει. Η κυρία Παρβάνοβα προσπαθήστε να τηρήσετε τα τέσσερα λεπτά, ώστε και τα υπόλοιπα ονόματα που ανέφερα προηγουμένως να προλάβουν τουλάχιστον να θέσουν ερωτήσεις. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Γκλένης για την ε, παρουσίασή της και ε, της έκθεσης και των τροπολογιών. Είναι μεγάλος ο αριθμός των τροπολογιών. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να συνεργαστούμε εκ των προτέρων πριν την πληροφορία για να εντοπίσουμε πιθανούς συμβιβασμούς και κείμενο, κείμενο το οποίο θα το υποστηρίξουμε όλοι. Πολλές τροπολογίες έχουν καλές προθέσεις και κανείς δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, ευημερία, την υγεία ε, των ασθενών. Νομίζω ότι συμφωνούμε γενικά με τις ε, βασικές διατάξεις του κειμένου. Οι αρχές είναι ε, σημαντικές. Ας μην προβούμε σε πολλές καλοπιστικές απλώς τροπολογίες οι οποίες δύσκολα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε. Όχι επειδή ε, είναι περιττές, ε, όχι επειδή είναι αβάσιμες μάλλον, αλλά επειδή δεν είναι καλές για την οικονομία του λόγου. Για τις επιτροπές διοντολογίας θα πρέπει να, τις, να βελτιώσουμε το το κείμενο, όλοι συμφωνούμε και η Κομισιόν ότι η αρχή θα πρέπει να είναι ότι καμία δοκιμή, κλινική δοκιμή δεν θα πρέπει να εγκρίνεται, να ξεκινάει χωρίς ε, σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Δεοντολογίας σε εθνικό επίπεδο. Οι προτάσει της ηγέτριας είναι ένα, μια, ένα καλό πρώτο βήμα, ας, μην, ας αποφύγουμε μάλλον τις επαναλήψεις. Ε, άλλωστε, έχουμε και την αρχή τη επικοικότητα. Οι ορισμένε τροπολογίε παραβιάζουν την αρχή αυτή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ρόλο των επιτροπών διοντολογία. Το καλύτερο είναι να εστιαστούμε στο τι μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον κανονισμό και να εμπιστευτούμε περισσότερο τις Εθνικές Επιτροπές Διοντολογίας. Ε, και εγώ και άλλοι έχουμε προτείνει τροπολογίες που θα λάβουν υπόψη την ιδιαιτερότητα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων στην αξιολόγηση της υποχρέωσης ε, κλινικών δοκιμών. Όμως προσοχή ε, να μην υπερβάλλουμε και καταστήσουμε τις κλινικές δοκιμές ανέφικτες για, για τα ευάλωτα άτομα ιδιαίτερα να μην δημιουργήσουμε εμπόδια στην ανάπτυξη φαρμάκων, ενώ όταν μιλούμε για προστασία παιδιών ή ευάλωτων ομάδων, ατόμων με αναπηρίες ή ειδικέ ε, ανάγκες, ε, ε, ψυχικά προβλήματα κλπ. Έχω υποβάλει τροπολογίες και για την διάταξη που αφορά την ε, ασφάλεια και την εκθέσεις ε, ανεπιθύμητων παρενεργειών ε, για τις δοκιμές για φάρμακα που έχουν ήδη εγκριθεί ζητούμε να επιβληθεί υποχρέωση έκθεση στην, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια θέλουμε, πρέπει να αναρωτηθούμε το εξής τι θέλουμε να κάνουμε δημόσιο και για ποιο λόγο. Πότε θα πρέπει να δημοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες και πώς. Έχουμε διάφορες αναλεκτικές λύσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, την ε, περίληψη, ε, και την, μπορούμε δηλαδή να δημοσιεύουμε μόνο μια περίληψη ή τα συνολικά στοιχεία. Νομίζω πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε μια ισορροπία. Η πρότασή μου είναι πριν την ε, άδεια για την εμπορία να δημοσιεύεται μια σύνοψη και μετά την αδειοδότηση να δημοσιεύεται η κλινική, τα, να δημοσιεύεται τα πόρισμα της κλινικής δοκιμής. Από το 2010 ε, ήδη εφαρμόζεται ένα παρόμοιο σύστημα. Ευχαριστώ. Η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ. Πρώτα να ευχαριστήσω την Γκλένις για την ε, θαυμάσια εκθεσή της και επειδή συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τα όσα λέχθηκαν ήδη, θα πω το Ανακάλυψα ίσως κάπως καθυστερημένα ότι πολύ λίγα μόνο φάρμακα περνούν από κύκλους κλινικών δοκιμασιών που τελικώς καταλήγουν σε έγκριση. Πολλά φάρμακα τα οποία περνούν από κλινικές δοκιμασίες ήδη είναι εγκεκριμένα. Έχουν επομένως ένα πλεονέκτημα. Άρα, δεν μιλούμε εδώ για τη δημιουργία νέων ρηξικέλευτων φαρμάκων. Εκεί λοιπόν που είναι απαραίτητο θα πρέπει να γίνεται αυτή η διαδικασία και εκεί αυτή θα πρέπει να διέπεται από διαφάνεια και μετά από την έγκριση. Αλλά για φάρμακα τα οποία ήδη είναι εγκεκριμένα και καμιά φορά ίσως τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα και μετά απευθύνονται στους γιατρούς και, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ή αλλιώς. Πάντως υπάρχουν και πολλά σκάνδαλα που έχουν σημειωθεί και γνωρίζουμε ότι δεν δημοσιεύονται πάντα τα αρνητικά ε, πορίσματα των ερευνών. Όπως για παράδειγμα το σκάνδαλο της ΡΟΣ που τήρησε μυστικό το ότι τα πειράματα που έκανε είναι ότι Εάν είχαν δώσει παρασεταμόλ, αυτό θα είχε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα όπως το τάμιφλου. Και ξοδεύτηκαν δισεκατομμύρια ευρώ λόγω της ε, γρήπης των πουλερικών, λόγω της γρήπης των χείρων. Φανταστείτε, αν υπήρχε υποχρέωση να δημοσιεύονται όλα τα συμπεράσματα των κλινικών ερευνών, θα είχαν αποφευθεί τέτοια σκάνδαλα. Όλα αυτά έχουν ωστόσο αρνητικέ συνέπειε γιατί κινδυνεύουν άλλοι ασθενεί για του οποίου δεν μπορούν να δαπανηθούν τα χρήματα αυτά. Θα γίνουν άραγε πιο έντιμε οι βιομηχανίε εάν υποχρεούνται να δημοσιεύουν όλα τα στοιχεία. Πάντως πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια να υποβάλλονται οι εκθέσεις, να, υποχρεωτικά οι εκθέσεις των κλινικών ερευνών. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα, θα υπάρχει δυνατότητα να ελέγχονται τα πορίσματα αυτά και δεν θα μπορεί η βιομηχανία να λέει ότι αυτά είναι δύσκολα. Δεν είναι δύσκολότερα ή περιπλοκότερα. Εφόσον υπάρχουν τα δεδομένα από τις κλινικές έρευνες, πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά. γιατί να προστατεύουμε τα οικονομικά συμφέροντα της βιομηχανίας σε βάρος των ασθενών. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ούτε θα το καταλάβουν και οι ψηφοφόροι, ούτε οι δικοί σας, ότι δηλαδή η Επιτροπή Περιβάλλοντος βάζει τέτοιε προτεραιότητε. Από την άλλη μεριά υπάρχουν βιομηχανίες οι οποίες θέλουν να είναι εντάξει, θέλουν να προστατεύσουν τα συμφέροντα των ασθενών. Και αυτές οι βιομηχανίες θα έχουν τότε καλύτερες, θετικότερες προοπτικές, διότι θα είναι πιο ισότιμοι οι όροι ανταγωνισμού εάν, και τότε θα υποφεληθούν οι έντιμες βιομηχανίες. Ελπίζω λοιπόν ότι με κοινή προσπάθεια θα μπορέσουμε να βάλουμε τον ασθενή στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Ο κύριος Σάμπερνοχ. Τέσσερα λεπτά κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, παρακολουθήσαμε τη συζήτηση μέχρι τώρα. Επιτρέψτε μου να σου κάνω εγώ ορισμένα ας πούμε πρόσθετα σχόλια. Ναι, η νομοθεσία είναι σημαντική γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε την ποιότητα την ποιότητα ζωής και την ουσία των ερευνών, των κλινικών ερευνών. Θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Θέλουμε όμως να έχουμε και ρωμαλαία δεδομένα, αξιόπιστα δεδομένα από τις κλινικές έρευνες. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Εγώ ανέφερα συχνά σήμερα την επικουρικότητα. Στη συγκεκριμένη πρόταση πιστεύω ότι κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε μια ορθή ισορροπία για το ποια πράγματα αποφασίζονται στο εθνικό επίπεδο, δηλαδή την ενήμερη συνένεση ε, σχετικά με τις αποζημιώσεις, τον τρόπο πρόσληψης των ε, υποκειμένων στις ε, κλινικές έρευνες. Νομίζω ότι αυτά μπορούν να ρυθμιστούν και σε υπερεθνικό επίπεδο. Εγώ συζήτησα τη συζήτηση αυτή και για τον εθνικό μας οργανισμό. Συχνά οι άνθρωποι είναι λίγο αρνητικοί, ιδίως όσον αφορά την σύντμηση των προθεσμιών των κλινικών ερευνών. Κυρίως τον χρόνο εγκρίσεως. Αυτό προφανώς δεν είναι πρόβλημα μόνο της δικής μου χώρας, γι' αυτό και πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Επίσης η ενήμερη συνένεση, διότι το υποκείμενο ο ασθενής Δηλαδή, όταν είστε ασθενείς και γίνεται υποκείμενο της κλινικής έρευνας, Αυτό, ασφαλώς αυτό αποτελεί παρέμβαση στην προσωπική σας, προσωπική ζωή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι πλήρως ενήμερο, ότι έχει ενημερωθεί από ειδικό που μπορεί να το εξηγήσει και όλους τους ενδεχομένους κινδύνους. Πρέπει να μιλήσουμε επίσης και τους, ε, για τις περιπτώσεις των αναπήρων. όπου για, για τις κατηγορίες αυτές η ενήμερη συνένεση είναι κέρια σημασίας. Η λήψη των αποφάσεων πρέπει να γίνεται σε, μία, σε ένα επίπεδο. Πρέπει να είναι ένα επίπεδο αρμόδιο για την λήψη της αποφάσεως. Επομένως, ο φορέας αυτός που θα οριστεί πρέπει να γίνεται από τη χώρα μέλος όπου θα διεξαχθεί η κλινική έρευνα. Αυτό πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο διοικητικά, τις διοικητικές πτυχές αλλά και τις διοντολογικές. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Ενιαία βάση δεδομένων. Μια ενιαία πύλη δηλαδή. Ιδίως σε ορισμένες χώρες μέλη, πόσα βλέπω εγώ από την εμπειρία μου δηλαδή, η κατάσταση είναι κάπως αβέβαιη. Η χώρα μέλος που συντάσσει την έκθεση πρέπει να διαρωτηθεί αν θα περιλάβει όλες τις απόψεις των άλλων χωρών μελών. Και αν είναι σε θέση να το πράξουν αυτό έγκαιρα. Όταν αρχίσαμε αυτή τη συζήτηση για τις κλινικές ε, δοκιμές, η γνώμη μας ήταν ότι η πρόταση της Επιτροπής ε, ήταν κάκιστη και θα ήταν καλύτερα να παραμείνουμε με την τρέχουσα οδηγία παρά να την αντικαταστήσουμε με μία πρόταση σαν ε, εκείνη της Κομισιόν. Θυμάμαι για παράδειγμα εδώ τη γνωμοδότηση της ομάδας μου αλλά και άλλων ε, ε, ομάδων με βάση τη γνωμοδότηση της ε, Παγκόσμιας Οργάνωσης Ιατρών που θεωρούσε ότι παραβιάζουμε τις δηλώσεις του Ελσίνκη και παραβιάζει κάθε επιτροπή δεοντολογίας κάθε δεδομένο περί Επιτροπής Δεοντολογίας ως προς τις ε, κλινικές δοκιμές. Φαίνεται λοιπόν ότι ξαναθέτουμε τα πράγματα στη σωστή τους ε, διάσταση με την πληθώρα τροπολογιών ως προς τις Επιτροπές ε, Δεοντολογίας. Θεωρούμε λοιπόν ως Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για απλούστευση της διαδικασίας. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι πολλά μέλη αυτής της Επιτροπής από πολλές πολιτικές ομάδες υπέβαλαν κοινέ τροπολογίες για αυτό το θέμα όπως και για πολλά άλλα. Οι τροπολογίες αυτές θα πρέπει να εγκριθούν όταν φτάσει η στιγμή της ε, ψηφοφορίας. Επίσης, η έκθεση της Γκλένης βελτιώνει την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί μια καλή βάση εργασίας. Ως προς τις γνωμοδοτήσεις και τις αρχές δεοντολογίας θεωρούμε ότι θα πρέπει να φορούν όλα τα εξελιγμένα κράτη-μέλη και θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα του opt-out για ένα κράτος μέλος, μέλος με βάση ε, ως προς μάλλον θέματα δεοντολογίας. Σε σχέση με την συνένεση, τη διαδικασία συνένεσης, αφορά και τις κλινικές δοκιμές και εντάσσεται στη θεμελιώδη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλούσαμε για ε, διαδικασίας διάγνωσης in vitro και ο Πέτερ Λίζε αναφέρθηκε σε αυτό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τα ε, δικαιώματα των πιο ευάλωτων κατηγοριών, ιδιαίτερα για τη συμμετοχή στις κλινικές δοκιμές. Επίσης, θεωρούμε ότι ε, ο ιστότοπος είναι ύψης της σημασίας για να διασφαλίσουμε και τη διαφάνεια και τα αποτελέσματα. Θα μπορούσαμε να έχουμε εκθέσεις λεπτομεριακές ή συνόψεις σε σχέση με δοκιμές, αποτελέσματα αυτών αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε ποιες είναι οι δοκιμές που οδήγησαν σε θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα ή δεν οδήγησαν σε αποτελέσματα. Πιστεύω ότι έχουμε μία καλή βάση για τροπολογία συμβιβασμού που μπορούν να μετατρέψουν την αρχική πρόταση σε ένα νομοθετικό κείμενο που να είναι το σωστό και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ασθενών και των πολιτών γενικότερα. Ευχαριστώ. Ακολουθούν τώρα οι λοιποί συνάδελφοι με τρία λεπτά για τον καθένα. Έχουμε περίπου μία ώρα στη διάθεσή μας. Ξαναλέω τα ονόματα. Kukovic, Hittner und Rossi. Habe ich noch jemanden vergessen? Μήπως κάποιος δεν άκουσε το όνομα του. Ο κύριος Κουμουτσάκος. Κύριε Γκροστέτ, πρώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα τρία λεπτά. Είναι αλήθεια ότι η πρόταση Κομισιόν ήταν καλή, η έκθεση είναι καλή. Ε, Ας μην επιστρέψουμε στις αδυναμίες της προηγούμενης οδηγίας. Ε, σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Διοντολογίας ε, συμφωνώ να αναφερθεί ρητά ε, το όνομα και ο ρόλος της, όμως το κείμενο δεν χρειάζεται να ορίσει το πεδίο εφαρμογής και τις αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Διοντολογίας. Είναι θέμα επιτροπολογίας. Συμφωνώ με την αναλογική προσέγγιση του κινδύνου, επιτρέπει την μείωση του διοικητικού άχθους για τις ε, δοκιμές ε, χαμηλής, ε, χαμηλού κινδύνου σε ό,τι αφορά την πρόσβαση πληροφορίες ε, μάλλον σε ό,τι αφορά την ε, απουσία ε, αποδοχής ε, έγκρισης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είναι καλό να θεωρείται ως σιωπηρή έγκριση. Σε ό,τι αφορά την διαφάνεια θα πρέπει να είναι ισορροπημένη, να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των μερών, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής έρευνας. Συνεπώς, θα πρέπει να δώσουμε σημασία στο timing των δημοσιεύσεων και στο περιεχόμενό τους. Σε ό,τι αφορά τη βάση δεδομένων που θα επιτρέπει να δίνονται στο κοινό πληροφορίε, πρέπει οι πληροφορίε αυτέ να είναι αξιόπιστε, να γίνονται σεβαστή και πάλι η ανταγωνιστικότητα. Οι δημόσιε πληροφορίε θα πρέπει να προστατεύουν τα απόρριτα προσωπικά δεδομένα αλλά και τα εμπορικά ε, ε, μυστικά ε, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προκειμένου να αποφύγουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό η ε, προθεσμία δημοσίευσης είναι πολύ σημαντική για να αποφύγουμε ακριβώ τον αθέμητο ανταγωνισμό που θα μπορούσε ασφαλώ να βλάψει την ανταγωνιστικότητα τη ιατρική ευρωπαϊκή έρευνα. Έχουμε υποβάλει κάποιε τροπολογίε μαζί με συναδέλφου για αυτό το θέμα. Ε, επιμένω επίσης ένα τελευταίο ζήτημα. Πρόκειται για τι σπάνιε ή πολύ σπάνιε ασθένειε Και εδώ έχω υποβάλει τροπολογίε γιατί θεωρώ πω είναι δύσκολο να γίνει κλινική δοκιμή που να λέω σε, για τέτοιου είδους ασθένειες γιατί συνδέεται με ένα πολύ μικρό αριθμό ασθενών για κάθε ασθένεια και ε, με μια μεγάλη γεωγραφική έκταση. Συνεπώς ε, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη η σπάνη της ασθένειας ε, το πόσο σπάνια δηλαδή είναι μια ασθένεια σε αυτές τις διατάξεις. Έχω υποβάλει συγκεκριμένες ε, τροπολογίες μαζί με άλλους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την κυρία Βίλμοντ καθώς και τον Φιλίπ Ζουβάν που είναι ο σκιώδης ηγητής του Λαϊκού Κόμματος. Εξ ονόματος κύριου Ζουβάν, ο οποίος βεβαίως είχε μόνο τέσσερα λεπτά στη διάθεσή του, θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν όντως η ψηφοφορία πρέπει να γίνει τον Απρίλιο, διότι έχουμε πολλές τροπολογίες αυτό βέβαια θα συζητηθεί μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Ο σκιώδης εισηγητής του Λαϊκού Κόμματο, κ. Ζουβά, ωστόσο, προτείνει να διαθέσουμε σε αυτού περισσότερο χρόνο. Η πρόταση τη Κομισιόν συνεπάγεται ορισμένα πλεονεκτήματα, λιγότερη γραφειοκρατία και βεβαίω και ζητεί περισσότερη διαφάνεια. Μπορεί να βελτιώσει κανεί την πρόταση τη Κομισιόν. Πάντω είναι ήδη πλεονέκτημα το γεγονό ότι η ίδια η Κομισιόν τα προτείνει αυτά. Θα πω στην κυρία Άουκεν ότι όταν γίνεται έρευνα για υφιστάμενες ουσίες δεν σημαίνει αυτό ότι έχει ταπεινά κίνητρα η βιομηχανία. Καμιά φορά είναι απαραίτητο ανεξάρτητοι ερευνητές για να εξετάσουν για παράδειγμα στην ογκολογία χρειάζονται οι έρευνες εφαρμογής για να εξεταστεί αν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει ορισμένους καρκίνους με λιγότερη χημειοθεραπεία. Άρα δεν είναι τα πράγματα άσπρα ή μαύρα. Μπορεί να υποστηρίξει κανείς ορισμένα από αυτά που ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, στο τέλος, για να μπορέσει να υπερψηφιστεί το κείμενο, χρειαζόμαστε επιγόντως αλλαγές σε τρεις σημαντικούς τομείς. Όπως είναι η πρόταση αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορούσα ούτε και εγώ να την υπερψηφίσω. Ως πρώτον, λοιπόν, θα έλθω σε αυτό που είπε ο κ. Σάβρενοχ, το πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί να συνενέσει το ίδιο, για παράδειγμα παιδιά ή διανοητικός ανάπηρη Είχαμε μια σχετική συζήτηση με την Κομισιόν την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε. Μας είπε ο κύριος Ρίγης ο Διευθυντής, ότι είναι η ίδια, το ίδιο κείμενο της οδηγίας του 2001. Ωστόσο καθίσαμε και το εξετάσαμε λέξη προς λέξη και είδαμε ότι δεν είναι το ίδιο κείμενο μαζί με την Κομισιόν. Αυτό πρέπει να τροποποιηθεί, θα πρέπει να είναι το ίδιο κείμενο του 2001 μαζί με πολλούς συναδέλφους πολλών χωρών μελών αλλά και πολλών πολιτικών ομάδων έχουμε συνεργαστεί για να καταθέσουμε τροπολογίες και παρακαλώ να τις στηρίξετε. Πρόκειται συνολικά για 7 τροπολογίες που έχουν ως σκοπό να επαναφέρουν την κατάσταση του 2001. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε για παιδιά ή για διανετικός αναπήρους να ισχύσουν λιγότερο αυστηροί κανόνες από την οδηγία του 2001. Τώρα, η σχέση της αρμόδιας επιτσουσίας χώρας και οι άλλες συναρμόδιες χώρες. Στην πρόταση της Επιτροπής η πρώτη αρμόδια χώρα έχει πολύ ισχυρό ρόλο. Εάν οι άλλες αρμόδιες χώρες θέλουν να συμβάλλουν στο αποτέλεσμα με την τεχνογνωσία τους δεν λαμβάνονται τόσο πολύ υπόψη. Εγώ δεν θέλω να έχουμε μόνο το λεγόμενο opt-out. Το Συμβούλιο θα πει κατά πάσα πιθανότητα 100% opt-out. Θα έχουμε πάλι όμως την αταραχή ότι τελικά δεν θα μπορούν να γίνουν ευρωπαϊκές κλινικές δοκιμές. Μπορώ να υποστηρίξω βεβαίω κατά τα άλλα τα περί δεοντολογικών επιτροπών και χωρί θετική ψήφο τη Δεοντολογική Επιτροπή δεν θα πρέπει να αρχίζει η κλινική έρευνα. Ευχαριστώ. Πετελίζε η κυρία Εστρέλα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Γκλένης για την εξαιρετική της ε, εργασία ε, σε σχέση με την ε, αρχική πρόταση της Κομισιόν. Εγώ μαζί με άλλους συναδέλφους υποβάλαμε τροπολογίες σε σχέση με ορισμένες ανησυχίες μας μετά από ανάλυση του εγγραφού. Μας απασχολεί η παράληψη της δράσης των Επιτροπών Δεοντολογίας και η εποπτεία της ευημερία του ασθενούς και επίσης ότι έχουμε προθεσμίες που είναι ε, πολύ αυστηρές σε σχέση με τις διαδικασίες δοκιμών. Σε σχέση με τις προθεσμίες αυτές, ίσως χρειάζεται και μια διαδικασία ή μια αυτοματοποιημένη αδειοδότηση για τις κλινικές δοκιμές. Θα πρέπει λοιπόν οι αρμόδιες αρχές να μπορέσουν να αναθεωρήσουν τους φακέλους αδειοδότησης. Επίσης, οι φορείς κλινικών δοκιμών θα πρέπει να επιλέξουν το κράτος μέλος που επιθυμούν, έτσι ώστε να μην επιλέγει κανείς ό,τι επιθυμεί από κάθε κράτος μέλος το οποίο έχει μία πιο χαλαρή πολιτική. Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας αδειοδότησης η προθεσμία έγκρισης και αδειοδότησης αφορά ε, μία προθεσμία έξι μερών που είναι πολύ στενή προθεσμία γιατί χρειάζεται μία μελέτη του πρωτόκολλου έρευνας, η οποία να είναι λεπτομεριακή. Γι' αυτό οι κλινικές δοκιμές θα πρέπει να είναι προσβάσιμες στο κοινό, είτε έχουν θετικό είτε αρνητικό αντίκτυπο. Αυτό δεν σημαίνει επιπρόσθετη ε, γραφειοκρατία, ούτε θέτει ένα αμφιβόλο τα προσωπικά δεδομένα, ούτε το ε, καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας. Γιατί πρέπει να γίνει μία επαναθεώρηση της όλης διαδικασίας και θα πρέπει να θεωρηθεί νέα διαδικασία χωρίς να λάβουμε υπόψη το ιστορικό, κάτι το οποίο θα βοηθούσε πολύ στην αξιολόγηση. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθεί για λόγους διαφάνειας και για να μην υπάρχει επιπρόσθετη γραφειοκρατία στη διαδικασία αδειοδότησης. Αυτές είναι οι ανησυχίες μας ε, τις οποίες εκφράζουμε σε συγκεκριμένες τροπολογίες που έχουμε υποβάλει. Merci, merci Monsieur Président. Moi, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει κυρία Ριβασί. Ευχαριστώ την κυρία Βουέλμοτ. Ε, με την έκθεσή της βελτιώνει πολύ την πρόταση της Κομισιόν. Θέλω να υπογραμμίσω τρία ζητήματα. Όλοι συμφωνούμε, νομίζω, ε, για την Επιτροπή Διοντολογίας ε, που είχε αφαιρεθεί. Χρειάζεται όμως να εναρμονιστούν οι Επιτροπές Διοντολογίας, διότι αν δημιουργηθούν προβλήματα μεταξύ κρατών μελών, αν οι επιτροπές διοντολογίας δημιουργούν εμπόδια, μάλλον αν υπάρχουν εμπόδια στην διενέργεια περισσότερων ε, κλινικών δοκιμών στην Ευρώπη, ίσως αυτό να οφείλεται και στη λειτουργία των επιτροπών διοντολογίας. Ε, το, ε, χρειάζεται να εναρμονιστούν τα πρωτόκολλα, οι πληροφορίε για τους ασθενείς κλπ. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο και οι χορηγοί θα ε, έχουν, ε, οι ανάδοχοι μάλλον, θα έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Ε, δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι η διαφάνεια. Ακούω τους συναδέλφους και όλοι λένε είμαστε υπέρ διαφάνειας, αλλά, αλλά αυτό το αλλά θα πρέπει να το διαγράψουμε. Η διαφάνεια των κλινικών δοκιμών σημαίνει πρόσβαση. Πρόσβαση όχι μόνο σε μια σύνοψη, αλλά στο σύνολο των δεδομένων γίνεται λόγος για μεταναλύσεις. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μετααναλύσεις. Γιατί εξετάζουν τα δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί και <clears throat> διαπιστώνουν αν τα αποτελέσματα είναι θετικά, αρνητικά ή ε, ανεπαρκή για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Το ταμιφλού, θυμάστε, πουλήθηκαν, που, πουλιότανε ε, κατά εκατομμύρια χωρίς να υπάρχουν οριστικές μελέτες για την αποτελεσματικότητά του. Εγώ είμαι υπέρ της πλήρους διαφάνειας και μου μιλάνε για το εμπορικό απόρριτο. Όχι. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, όχι το εμπορικό απόρριτο. Καμία σχέση με εμπορικά δεδομένα. το εργαστήριο Abbott ε, ε, προσέφυγε εναντίον της, ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων γιατί δημοσίευσε στοιχεία, δεδομένα για φάρμακα. Εμείς θα πρέπει να την υπερασπιστούμε και να υπερασπιστούμε τη διαφάνεια με δημοσίευση των στοιχείων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας. Εμείς θα πρέπει να πολεμήσουμε υπέρ της διάδοση αυτών των πληροφοριών. Μετά, η χαμηλή επέμβαση. Ε, ε, ε, δεν με βρίσκει πολύ σύμφωνη για τις... αυτός ο όρος. Θυμάστε την έκθεση Regulate για ε, αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται όχι για διαβήτη, για την κατανόηση του διαβήτη, αλλά για μείωση του βάρους, για απώλεια βάρους και δημιουργούσε προβλήματα με τις βαλβίδες. Ε, ε θεωρείται λοιπόν χαμηλής παρέμβασης, αλλά βλέπετε ότι δεν ήταν. Μάλλον θα πρέπει <clears throat> να γνωρίσουμε καλύτερα τον όρο να τον καταργήσουμε. Ε, ευχαριστώ κύριο Σπερέλιο. συγχαρητήρια στην κυρία Βουελμότ ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κριτήριο της ε, διαφάνειας. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί με τον εαυτό μας. Ε, ε, και θα πρέπει να είμαστε και ισορροπημένοι, αλλά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή των ασθενών και το δικαίωμα στην πνευματική ιδιοκτησία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως άλοθη ή ως προσχήματα για να μην γίνονται πλήρες ε, κλινικές δοκιμές ή να κυκλοφορούν φάρμακα τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί επαρκώς ή ακόμα και ε, ε, να γίνονται, να σκούνται πρακτικές κερδοσκοπίας. Συνεπώς, το κριτήριο που δίνει η κυρία Γουίλμα ότι είναι καλό, βελτιώνει την, πρόταση κομισιών. Έχω υποβάλει τροπολογίες για την, τις επιτροπές διοντολογίας. Πράγματι υπάρχει διαφορά ε, μεταξύ κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη, λειτουργία των επιτροπών αυτών. Η λύση της ε, Κομισιόν ήταν να βάλει κάτω από το χαλί το θέμα και να μην αναφερθεί σε αυτές τις επιτροπές. Δεν είναι η πιο σωστή προφανώς ε, λύση, η πιο σωστή προσέγγιση. Εμείς είμαστε εδώ για να νομοθετήσουμε και να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ε, δεν είναι εδώ να τον τσαγνοήσουμε ακόμα και αν δεν μπορούμε να εναρμονίσουμε τη λειτουργία τους. Οι, όλες οι κλικές δοκιμές θα πρέπει να αξιολογούνται από τέτοιες επιτροπές. Ε, σε ό,τι αφορά του ευάλωτου πληθυσμού, επίση έχω υποβάλει τροπολογίε. Ε, θα πρέπει να τη χάνουν ιδιαίτερη ε, προστασία. Θα, ε, σε ό,τι αφορά τα παιδιά, θα πρέπει όταν είναι περισσότερο, όταν έχουν και μεγαλύτερο των 10 να δίνουν την ενεπιγνώση σύμφωνη γνώμη τους δεν είναι όμως μόνο τα παιδιά, η ανάπηροι, ευάλωτα άτομα. Ε, υπάρχουν και άλλα άτομα όπως οι έγκυες γυναίκες, ή άτομα που λόγω της οικονομικής κατάστασης μπορούν να είναι ευάλωτα άτομα για μια συγκεκριμένη δοκιμή. Θα πρέπει και αυτό να αξιολογηθεί. Ειδικά στην, ε, σε μια οικονομική κατάσταση τόσο δύσκολη όσο η, σημερινή, όσο η σημερινή. Για όλα αυτά τα άτομα θα πρέπει να έχουμε ειδική μέρημνα. Χρειάζονται ειδική προστασία και δεν θα πρέπει να τα αγνοήσουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Κούκοβιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ονομάζομαι ε, Μαζέη Κούκοβιτς. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να προφέρετε το όνομά μου. Ε, τι με απασχολεί περισσότερο σε αυτή την έκθεση. Η γύρανση του πληθυσμού. Η πνευματική υγεία και άλλα παρεμφερή ζητήματα. Και ιδιαίτερα, ή επίσης μάλλον, η υγεία των παιδιών. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μία πολύ δύσκολη περίοδο επειδή γυράσκει η Ευρώπη μας. Συμφωνώ με τον κύριο Λίζε, ο οποίος θα ήθελε να αναβληθεί η ψηφοφορία αυτή για να έχουμε τη δυνατότητα να συντάξουμε καλύτερα και να ρυθμίσουμε καλύτερα ε, ορισμένα επιμέρους ζητήματα και εγώ θα πρέπει να αντιταχθώ σε αυτές τις στενές προθεσμίες, διότι αν θέλουμε οι επιτροπές δεοντολογίας να μπορέσουν να εκφραστούν, το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να λυθεί εν μία νυχτή. Και σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου θα προβαίνουμε σε σιωπηλές εγκρίσεις και που θα αποτελέσουν πάγια πρακτική. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε λίγο μεγαλύτερες ε, προθεσμίες. Αυτό δεν αποτελεί καλύτερη λύση. Όλοι όσοι ασχολούνται με θέματα δεοντολογίας γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν έχουμε ερευνητές και εμπειρογνώμονες που να υπαρκούν τουλάχιστον στην Ευρώπη και πολλές φορές πρέπει να προστρέξουμε σε εμπειρογνώμονες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να λήξει σε λίγες μέρες. Και εγώ έχω υποβάλει τροπολογίες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι ελοχεύει κίνδυνος φυσικής και ψυχικής υγείας όταν μιλάμε για κλινικές δοκιμές. Είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να τονιστεί επαρκώς και ελπίζω να υποστηρίξετε τις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ κυρία Μασέη Κούκοβιτς. Σας υπόσχομαι ότι θα ασκηθώ και θα βελτιώνομαι από συνεδρία σε συνεδρία. Η κυρία Χίπνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή και την Κομισιόν, την Κομισιόν εννοώ, για το έγγραφο που μας υπέβαλε, που είναι τόσο σημαντικό για μεγάλο αριθμό πολιτών. Μιλούμε για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εισάγει τροποποιημένες διαδικασίες για τις κλινικές έρευνες. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, γιατί για πρώτη φορά κάνουμε προσπάθεια εναρμόνισης όλης της διαδικασίας με μια ενιαία πύλη διαδικτύου που θα επιτρέπει την κατάθεση αιτήσεων για τις δοκιμές αυτές. Και αυτό θα συνδέεται με την βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα είναι λοιπόν ενιαία η διαδικασία και θα ελέγχεται από τις χώρες μέλη που μπορούν να υποφεληθούν και από την ε, συνεργασία ειδικών οργανισμών. Οι αξιολογήσεις των κλινικών ερευνών θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με δεοντολογικές αρχές, καθώς επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Κάθε χώρα μέλος θα έχει την δυνατότητα να ορίζει τις ιδιαίτερες διαδικασίες της, εφόσον βέβαια συμμορφώνεται με τις διεθνείς guidelines όσον αφορά την ανεξαρτησία των αξιολογητών. Σημαντικό είναι επίσης ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια των κλινικών δοκιμών, διότι κάθε αίτηση θα αξιολογείται από πρόσωπα ανεξάρτητα και που θα διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη. Επίσης, η δραστηριότητα αυτή διακρίνεται από την δραστηριότητα έκδοσης εγκρίσεων για την διεξαγωγή των κλινικών ερευνών, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να αισθάνονται ασφαλέστεροι εν τέλει. Και αυτό αναφέρεται πράγματι μέσα στο κείμενο, δηλαδή κάθε πρόσωπο που θα συμμετέχει στις κλινικές δοκιμές θα πρέπει να έχει δηλώσει την ενήμερη, την ε, ενήμερη συνένεσή του εκτός από την αντιμετώπιση κατεπιγουσών περιπτώσεων βέβαια. Αυτά όλα σε ένα ενίο κείμενο. Είχαμε βέβαια μέχρι τώρα α, σχετικές διατάξεις, ήταν όμως κάτι σπαρμένες. Θα θεσπιστούν και βέλτιες πρακτικές και για τη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης προβλέπεται και αποζημίωση, προβλέπεται αποζημίωση δηλαδή, στην περίπτωση που οι κλινικές έρευνες προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες στα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές. Ευχαριστώ. Ρώση. Ευχαριστώ. Ήμουν αφηρημένος, με συγχωρείτε. Καταρχήν ευχαριστώ την ε, κυρία Βίλμοτ, συμφωνώ μαζί της για μία φορά και έχω υποβάλει και τροπολογίες. Ελπίζω να μπορέσουμε να συντονιστούμε για τις ως προς 700 τροπολογίες που υποβάλαμε όλοι και να φτάσουμε σε μία σύμπνοια με τροπολογίες συμβιβασμού που θα βρούμε γιατί το θέμα είναι πολύ σημαντικό για να το παραβλέψουμε. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, μιλάμε για κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους και όποιος ασθενεί και υπόκειται ε, σε τέτοιες κλινικές δοκιμές θέλει να σώσει τη ζωή του, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν είναι πάντα δεδομένο. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν όλες οι κατηγορίες ασθενών ε, ε, και ιδιαίτερα οι φυσικά ή ψυχικά μη υγιείς ή εκείνοι τους οποίους πρέπει να αναλάβουν τα παιδιά τους. Θα πρέπει λοιπόν να εξεύρουμε μεθόδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να είμαστε αρκετά οργανωμένοι και συντονισμένοι. Μιλάμε για ευημερία και ασφάλεια των ασθενών που θα πρέπει να υπερδεσπόζουν οποιασδήποτε άλλη σκέψη. Νομίζω ότι το κείμενο της κυρίας Βίλμοτ θα μπορέσει να αποτελέσει μία βάση συμφωνίας και ελπίζω να φτάσουμε σε αίσιο πέρας ως προς τις 700 αρχικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κουμουτσάκος. Ζητώ συγγνώμη γιατί κάπως ε, δυσκολεύτηκα με την εκφορά του ονόματός σας. Υπάρχει κου στο επώνυμο, υπάρχει μια δυσκολία. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, το σχέδιο της έκθεσης γενικά κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Και ευχαριστούμε τη συνάδελφο για τη δουλειά που έχει κάνει παρουσιάζοντας το συγκεκριμένο κείμενο εργασίας. Θα μπορούσαν πολλά να υποθούν άλλα υποστρικτικά και άλλα ε, που θα εξέφραζαν ένα προβληματισμό. Εγώ θα εντοπίσω την παρέμβασή μου σε ένα μόνο σημείο που ε, προκαλεί, κατά την άποψή μου, έναν έντονο προβληματισμό. Και αυτό είναι το σημείο του άρθρου 73. Δηλαδή, το άρθρο εκείνο που προβλέπει ε, την δημιουργία εθνικών μηχανισμών αποζημίωσης. Σε αυτό το άρθρο λοιπόν προβλέπεται ότι ένας εθνικός μηχανισμός αποζημίωσης θα λειτουργεί σε όλα τα κράτη-μέλη για την αποκατάσταση τυχών ζημιάς που μπορεί να υποστεί κάποιος που συμμετέχει σε κλινικές δοκιμές. Η πρόταση εκ πρώτης όψεως κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Πολύ φοβάμαι όμως ότι στην πραγματικότητα δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει εξίσου προς όφελος όλων των ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το λέω διότι είναι ένα γεγονός στο οποίο, στο οποίο κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια ότι σε όλα τα κράτη-μέλη η εμπειρία και κυρίως η δυνατότητα να δημιουργηθούν τέτοιοι εθνικοί μηχανισμοί δεν είναι ίδια. Ειδικά σε περιόδους βαθιάς οικονομικής ύφεσης και πολύ μεγάλων πιέσεων για την μείωση των εξόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Επομένως, για να συνοψίσω, ούτε όλα τα κράτη έχουν την ίδια εμπειρία διαχείρισης και δημιουργίας τέτοιων ταμείων, αλλά ούτε όλα τα κράτη-μέλη, κυρίως λόγω της βαθιάς οικονομικής ύφεσης και της αρνητικής συγκυρίας, η οποία κανείς δεν μπορεί να ξέρει πόσο θα κρατήσει, αλλά και των πιέσεων στα έξοδα των ασφαλιστικών ταμείων κάνουν αυτή την πρόταση ενώ είναι γενικά καλή προβληματική. Η διαφορετική ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο θα λειτουργεί ένα εθνικό σύστημα θα έχει ως συνέπεια οι ασθενείς που συμμετέχουν στην ίδια διακρατική έρευνα να τη χάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης ανάλογα με τη χώρα που βρίσκονται. Έτσι το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ομάδων ασθενών δύο ταχυτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να παρακαλέσω και τους εισηγητές αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε ξανά πιο προσεκτικά το ζήτημα και να εξετάσουμε ορισμένες πιθανές αναλλακτικές λύσεις άμεσα πραγματοποιήσιμες. Ίσως, και το τονίζω αυτό, ίσως μια τέτοια λύση ήταν η δημιουργία ειδικών μηχανισμών αποζημίωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή κάθε κράτους μέλους. Οι μηχανισμοί αυτοί ευρω... Ε, ε, αποζημίωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούν να αξιοποιούν την εμπειρία και την δυνατότητα συνεργασίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, νομίζω ότι είναι ένα σημείο το οποίο χρήζει της προσοχής μας εάν δεν θέλουμε και πιστεύω ότι κανείς μέσα σε αυτή την αίθουσα δεν θέλει να δούμε να δημιουργούνται διαφορετικές ομάδες ασθενών διαφορετικών ταχυτήτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κουμουτσάκο. Θα ακούσουμε τώρα την Κομισιόν, εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας Καταναλωτών. Έχετε λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια κυρία Γουίλμοντ για την ποιότητα της εκθέσεώς της καθώς και τους και εισηγητές που συμμετέχουν σε αυτή τη σημαντική εργασία. Η παρέμβασή μου θα εστιαστεί σε δύο κυρίως θέματα που είναι κρίσιμα για τις προτάσεις και θεωρούνται θεμέλι λύθη της προτάσεως. Πρώτο, για την συμμετοχή των διοντολογικών επιτροπών και δεύτερο, για τα κοινά στάνταρ προστασίας των συμμετεχόντων στις κλινικές δοκιμές για το πρώτο θέμα, τον ρόλο των διοντολογικών επιτροπών. Αυτές είναι όργανα που αξιολογούν ορισμένες πτυχές των project κλινικών ερευνών. Με την ευκαιρία διευκρινίζουμε ότι ποτέ δεν ήταν στόχος της προτάσεως της Κομισιόν να καταργηθεί το έργο των διοντολογικών επιτροπών υπήρξε παρανόηση της προτάσεώς μας. Η πρότασή μας έχει ένα απλό στόχο, να διασφαλιστεί ότι το έργο των επιτροπών αυτών αποτελεί μέρος της διαδικασίας εγκρίσεως για την διεξαγωγή των κλινικών ερευνών σε διάφορες χώρες μέλη. Για να επιτευχθεί αυτό, δίνουμε μεγάλο περιθώριο στις χώρες μέλη να ιδρύσουν διοτολογικέ επιτροπές και να τις εντάξουν στο σύστημά τους. Εδώ θα σεβαστούμε τις παραδόσεις των χωρών μελών και τη σχετική τεχνογνωσία τους θα λάβουμε υπόψη προσεκτικά τις προτάσεις που ενδέχεται να συμβάλλουν στην διευκρίνηση της προσεγγίσεως αυτής. Τονίζω και πάλι ότι το έργο των δεντολογικών επιτροπών θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα της διαδικασίας της εγκρίσεως διεξαγωγής κλινικών ερευνών και όχι ξεχωριστή παράλληλη διαδικασία. Για το δεύτερο θέμα, κοινού κανόνες και επίπεδο προστασίας. Οι δύο βασικοί στόχοι της προτάσεως της Κομισιόν έχουν ως εξής. Πρώτον, να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο των υποκειμένων των κλινικών δοκιμών. Δεύτερο, ευθυγράμμιση ή ενοποίηση των κανόνων σε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε αποφασίσαμε να δώσουμε μορφή κανονισμού. Αν θέλουμε να έχουμε κοινή αξιολόγηση από πλευρά των χωρών μελών, θα πρέπει τότε οι χώρε μέλη να είμαστε βέβαιοι ότι εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια για την αξιολόγηση των κλινικών ερευνών. Ακόμα και αν είναι διαφορετικά τα κριτήρια, διότι αν είναι διαφορετικά τα κριτήρια δεν θα αποδώσει η κοινή αξιολόγηση. Γι' αυτό και το Κοινοβούλιο ζήτησε κανονισμό και όχι οδηγία και εισακούστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεσπίζοντας τα κριτήρια στην πρόταση, ακολουθήσαμε την υφιστάμενη οδηγία και είναι στην ουσία ταυτόσιμα τα κριτήρια. Αυτό είναι σωστό διότι οι κανόνες, σε τους κανόνες βασίζονται και τα διεθνή στάνταρτ και οι γραμμές. Θα ε, εξετάσουμε και τις τροπολογίες που θα βελτιώσουν τον κανόνα αυτό. Ωστόσο, είναι κρίσιμο για την ορθή λειτουργία του κανονισμού να διατηρηθεί ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα εφαρμόζεται στην έγκριση των κλινικών ερευνών. Και τέλος, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε. Πέρσι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, ο αριθμός των κλινικών ερευνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε και πάλι κατά 10%. Όλοι λοιπόν θα επωφεληθούν από αυτήν την νομοθεσία. Θα επωφεληθεί η Ευρώπη, θα επωφεληθούν οι ασθενείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τέλος, η εισηγήτρια η οποία έχει το δύσκολο καθήκον που αγγίζει τα όρια του τετραγωνισμού του κύκλου με διαδίτη και κανόνα να, να βάλει σε ένα ενίο σύνολο σε 700 τροπολογίες. Για διαδικαστικό θέμα, ε, γιατί δεν, ε, για το θέμα που έθεσα δεν υπήρξε καμία αντίδραση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα των ε, μηχανισμών ταμείων, των, ε, μηχανισμών αποζημίωσης. Ε, δεν υπόθηκε τίποτα. Η, ο της Κομισιόν ανέγνωσε κείμενο. Ίσως είναι σε θέση η Κομισιόν τώρα, γιατί έχουμε και τον απαιτούμενο χρόνο, να απαντήσει στο ερώτημα του συναδέλφου. Το θέμα αυτό σχετίζεται με τον εθνικό νόμο που διαφέρει από χώρα σε χώρα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο να ισχύσει παντού. Ε, οι διατάξεις διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και θεωρήσαμε ότι το σύστημα αυτό είναι σκόπιμο γιατί σε αυτή την περίπτωση θα είναι δύσκολη ε, η, εφαρμογή στα εθνικά συστήματα αν ορίσουμε ένα ευρωπαϊκό, ε, μια ευρωπαϊκή στάθμη του ζητήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ε, συζήτηση. Ήταν άκρος ενδιαφέρουσα Ξέρουμε ποιοι είναι οι τομείς που δημιουργούν διφορούμενα ως προς τις επιτροπές ε, δεοντολογίας. Η Επιτροπή δεν ήθελε να τις απορρίψει από αυτή τη διαδικασία ή να τις αποβάλει και όλες οι κλινικές δοκιμές θα υπόκεινται στην προγενέστερη συμφωνία των Επιτροπών Δεοντολογίας στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό πρότεινα να έχουμε μία πλατφόρμα όπου θα συναντώνται οι Επιτροπές Δεοντολογίας για να μιλήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις για τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά οι Επιτροπές Δεοντολογίας συμμετέχουν και στους δύο και στα δύο σκέλη της νομοθέτησης. Ως προς τη διαφάνεια είπα ότι υπάρχει διαφορά ως προς την άποψή μας για τη διαφάνεια. Μερικοί θέλουν όλα τα δεδομένα, άλλοι θέλουν σύνοψη. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ε, διαφοροποίησης και γι' αυτό προσπάθησα να φτάσω σε μία μέση οδό. Καθίσταται σαφής, σαφές το ζήτημα της εμπορικής, του εμπορικού απορρίτου, όπως είπε η Επιτροπή. Και αυτό αφορά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ως προς τις ευάλωτες ε, ομάδες, ε, είδαμε το κείμενο του 2001 και έχω προσθέσει και μία παράγραφο για τις ευάλωτες ομάδες. Θα το συζητήσουμε όμως. Αυτά τα ζητήματα μπορούν να συζητηθούν ως προς την χαμηλή παρέμβαση, την ε, κατηγορία της χαμηλής παρέμβασης, ορίζεται στην πρόταση της Επίτροπης και θα ήθελα να ρίξετε μια ματιά γιατί είναι σαφές τι σημαίνει χαμηλή παρέμβαση. Είναι ένα θέμα πολύ, μια σημαντική πτυχή της πρότασης, διότι αυτή η κατηγορία θα κάνει μεγάλη διαφορά για όσους εργάζονται στον τομέα. Η κυρία Γκροστέτ μίλησε για τις σπάνιες ασθένειες. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποτελέσουν απόλυτη προτεραιότητα. Συμφωνώ λοιπόν με όσα προείπατε και συμφωνώ με τον κύριο Ρώση, γιατί και αυτό συμφωνεί μαζί μου. Ως προς τα εθνικά συστήματα αποζημίωσης, νομίζω ότι πολλοί ανησυχούν χωρίς να ξέρουν γιατί μιλάμε. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανείς υπερβολικά. Σε ορισμένες χώρες λειτουργεί πολύ καλά αυτό το σχήμα, αλλά το κόστος ασφάλισης είναι πολύ υψηλό και οντιστάθμισμα πολύ χαμηλό αλλά γι' αυτό ακριβώς δεν γίνεται κατανοητός ο φόρτος από τους ανθρώπους, διότι αυτό έχει, έχει θυγεί πολλές φορές και ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε το δανέζικο πρότυπο, γιατί φαίνεται να είναι, άκρο, να είναι άκρος λειτουργικό. Οι μικρότερες χώρες ανησυχούν ιδιαίτερα. Αυτό μπορεί να μας απασχολήσει να το συζητήσουμε. Υπάρχει κοινό έδαφος και νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ καλούς συμβιβασμούς εάν το επιθυμούμε. θα μιλήσουμε με τους σκιώδεις για ενδεχόμενες τροπολογίες συμβιβασμού στο εγγύς μέλλον και ελπίζω πριν από το τέλος της θητείας να έχει λήξει το θέμα, να έχει ψηφιστεί. Ευχαριστώ κύριε, κύριε, Καλή επιτυχία. Όπως είπα είναι μια εργασία μαμούθ. Για την περαιτέρω διαδικασία προβλέπουμε στις 24-25 του μηνός εδώ, Απριλίου, Απριλίου διορθώνουμε, εδώ στην ε, Επιτροπή Συζήτηση θα πρέπει οι εισηγητές και οι σκιώδεις να συμφωνήσουν εάν θα ε, ζητήσουν κάποια αναβολή, ακόμη δεν έχω κανένα σχετικό στοιχείο. Θα γίνει η ψηφοφορία όπω λοιπόν, όπως είπα, 24-25 Απριλίου. Η συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια ακόμη δεν έχει καθοριστεί. Βέβαια θα εξεταστεί από την περαιτέρω πορεία αν θα υπάρξουν πολλέ συμβιβαστικέ τροπολογίε ή όχι και πώ θα χειριστεί το θέμα. Ω πρόεδρο τη επιτροπή, ωστόσο, θέλω να είναι εξασφαλισμένο ότι δεν θα καταλήξουμε στην Ολομέλεια με 700 τροπολογίε αλλά με όσο δυνατόν λιγότερες. Θέλω να το αποφύγω ως πρόεδρος να ξανά έχουμε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή των ε, γεωργικών. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Έχουμε έτσι ολοκληρώσει τη συζήτηση του θέματος 11 της ημερησίας διατάξεως και τώρα ερχόμαστε στην συζήτηση με τον Επίτροπο κύριο Ταγιάννη. Καθώς όμως έχουμε ολοκληρώσει την συζήτησή μας ένα δεκάλεπτο πριν από την ώρα που προβλέπετε να προσέλθει, διακόπτω για ένα δεκάλεπτο την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας και μόλις προσέλθει ο κύριος Ταγιάννη θα επαναληφθεί η συζήτηση και ο Κρίς Τέιβις μπορεί ήδη να καθίσει και να είναι έτοιμος. Σύντομη διακοπή. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως στις 17.30. Υπότιτλοι So, wir nehmen die Sitzung wieder auf nach einer kurzen Unterbrechung. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση μετά από τη σύντομη διακοπή καλωσορίζω εγκαρδίως τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιο για τις επιχειρήσεις εδώ στην ε, Επιτροπή μας. Το θέμα μας είναι ψυκτικά υγρά των air condition στα αυτοκίνητα. Έχουμε τη σχετική διαδικασία. Ο κύριος Σταλιάνη θα λάβει το λόγο το πολύ για 10 λεπτά για να μπορέσει να διεξαχθεί και συζήτηση. Πολλοί συναδελφοί μας έχουν ζητήσει το λόγο και επιθυμούν να συζητήσουν με τον Επίτροπο κύριο Ταγιάννη και βλέπω να σηκώνουν διάφοροι τις καρτέλες τους. Ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής λαμβάνει το λόγο. Κύριε Ταγιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ πριν ε, περάσω στην ε, ουσία του θέματος, το οποίο με απασχόλησε αρκετά τους προηγούμενους ε, μήνες, θα ήθελα να μιλήσω για την βιομηχανική πολιτική γενικότερα διότι και το θέμα του ψυκτικού υγρού εντάσσεται γενικότερα στη βιομηχανική μας ε, πολιτική που να είναι πιο πράσινη, να σέβεται το περιβάλλον και να επιτρέψει στην Ευρώπη να ε, διαβεί, να υπερβεί αυτή την ε, κρίση. Και εμείς θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να σταματήσουμε την παρακμή της βιομηχανίας και όπως γνωρίζετε, στις 10 Οκτωβρίου εγκρίναμε τη νέα στρατηγική της βιομηχανικής πολιτικής με στόχο να έχουμε ένα 20% του ΑΕΠ της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020 που να προέρχεται από τη βιομηχανία, από τη βιομηχανία μας. Είναι ε, ένας πολύ φιλόδοξος στόχος, αφορά ιδιαίτερα την ε, καινοτομία και οι νέες δημοσιονομικές προοπτικές που ελπίζω να ε, εγκριθούν θα μας οδηγήσουν από 54 σε 80 δις τα κονδύλια για την καινοτομία και την έρευνα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να εκπονήσουμε μια συντονισμένη στρατηγική. Ε, τα συμπεράσματα του, Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της προηγούμενης ε, εβδομάδας δείχνουν μια ε, μεταστροφή. Εδώ και πολλά χρόνια μιλούσαμε για μια χρηματοοικονομική πολιτική και πολιτική υπηρεσιών που αποτελούν πρωταρχικό μας μέλημα πλέον. Είναι ένα θέμα που απασχολεί και εσάς και γι' αυτό θα ήθελα να αρχίσω από την αυτοκινητοβιομηχανία. Πρόκειται για το πρόγραμμα CARS 2020. Εγκρίναμε το Νοέμβριο, όπως γνωρίζετε, αυτό το πρόγραμμα, το οποίο όμως θα πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένα μέτρα. Καταρχήν θα πρέπει να υποστηρίξουμε την καινοτομία, και ελπίζω ότι θα φτάσουμε στον διπλασιασμό των κονδυλίων για την καινοτομία και το πράσινο αυτοκίνητο μέσα στα πλαίσια του ορίζοντα 2020, δηλαδή να περάσουμε σε 2 δις ευρώ από ένα θα πρέπει να μας απασχολήσει και μια εμπορική πολιτική που να μην είναι και τόσο αφελής. Εδώ λαμβάνω υπόψη και τις διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία και πριν από την υπογραφή θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχουν αρνητικές κυρώσεις για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Θα πρέπει να δώσουμε όθηση και, στη νέα μας, και στις νέες μας τεχνολογίες χωρίς επιπλέον άχθος. Άρα το ΚΑΡΣ 2020 αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση στην Ευρώπη μεταξύ κατασκευαστών, προμηθευτών και πελατών. Πολλές φορές δεν υπάρχει επαρκής καινοτομία. Γι' αυτό η αποδοτική στρατηγική CARS 2020 αποτελεί μια προσπάθεια συντονισμού μεταξύ βιομηχανίας, συνδικάτων, των εθνικών αρχών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Θα σας ορίσω τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η Επιτροπή. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που έγινε με τη Χαλιβουργία 35 χρόνια πριν με το επωνομαζόμενο πρόγραμμα Νταβινιών, το οποίο όρισε την επαναδιάρθρωση της Χαλιβουργίας με βάση ποσοστώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αυτοκίνητο βιομηχανία δεν υπάρχουν νομικά μέσα ούτε και οι οικονομικοί όροι και προϋποθέσεις. Η Επιτροπή μπορεί να προλάβει άδικες ε, παραβάσεις και στρεβλώσεις. Το σχέδιο ΚΑΡΣ 2020 προβάλλει συγκεκριμένα μέτρα για να λάβουν υπόψη τις αλλαγές του ΟΝΤΟΜΕ. Έχουμε προβεί στη σύσταση Task Force για να ε, δούμε περιπτώσεις κλεισίματος ε, μονάδων και μετά από αίτημα της βελγικής κυβέρνησης έχουμε αρχίσει τις διαδικασίες της Task Force για, την, ε, για το κλείσιμο του εργοστασίου Ford στη Γκένκ. Θα χρησιμοποιήσουμε κοινοτικά και ευρωπαϊκά κονδύλια για ε, επαναδιαπραγμάτευση. Με τον Επίτροπο Άντορ ορίζουμε τις βέλτιστες πρακτικές για να μπορέσουμε να επαναδιαρθρώσουμε τον τομέα. Σε σχέση με τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και όπως ζήτησε και ο πρόεδρος Γκρότε θα ήθελα να σας μιλήσω για την οδηγία 2006 κάθετο 40 για τις μονάδες κλιματισμού των οχημάτων που αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ μόν πριν από έξι μήνες. Από την 1η Πρώτου 2011 τα αυτοκίνητα θα πρέπει να φέρουν ένα συγκεκριμένο ψυκτικό υγρό το οποίο θα έχει δυναμικό αύξηση της θερμοκρασίας κατώτερο των 150 μονάδων. Και έτσι θα μειώσουμε και ε, τα αέρια θερμοκηπίου όπως ορίζει η οδηγία. Δεν πρόκειται για... παρά για το γεγονός ότι η αύξηση βιομηχανία θα πρέπει να, να χρησιμοποιεί το ψυκτικό υγρό HFO 1234YF από το 9 και μετά. Όπως γνωρίζετε, οι αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποιούν αυτό το υγρό στον κλιματισμό αυτοκινήτου, διότι έτσι μπορεί να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση ως προς τις επισκευές, την επισκευή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό η Επιτροπή ζήτησε και προσωρινή εξαίρεση για την εφαρμογή της οδηγίας. Με βάση λοιπόν τις ε, έκτακτες συνθήκες, επειδή υπήρχε σπάνης αυτού του ψυκτικού υγρού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 12 δεν θα ξεκινούσε διαδικασίες επί παραβάση στην περίπτωση που δεν υπήρχε συμμόρφωση κατά την πιστοποίηση των οχημάτων που έχουν κατασκευαστεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2012. Όταν συναντηθήκαμε, σας είπα ότι δεν θα δεχτώ νέες παρατάσεις και από την 1η Ιανουαρίου του 2013 η οδηγία θα εφαρμοστεί πλήρως σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω αυτή μου τη θέση όπως σας την εξέφρασα έξι μήνες πριν. Δεν έγινε καμία παράταση, καμία εξαίρεση, άρα η οδηγία έχει τεθεί σε ισχύ από την πρώτη χρησιμοποίηση αυτού του αερίου δεν χρησιμοποιείται πλέον στα οχήματα και εάν γίνει κάτι τέτοιο τότε οι κατασκευαστές παραβαίνουν το νόμο. Ζητήσαμε πληροφορίες από τα κράτη-μέλη και παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις κατά την εφαρμογή κατά εφαρμογή της οδηγίας σε σχέση με θέματα ασφαλείας για τη χρήση του νέου αερίου γιατί έγινε λόγος για την εφαρμογή της οδηγίας σε ορισμένες χώρες, θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οριστικές αξιολογήσεις για να μπορέσουμε, τις οποίες να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε. Η Επιτροπή θεωρεί την ασφάλεια των πολιτών άμεση προτεραιότητα και, θα, και παρακολουθούμε το ζήτημα εκ του σύνεγγης. Άρα δεν μπορούν να τεθούν στην αγορά ε, προϊόντα που δεν συμμορφούνται προς αυτές τις ε, προδιαγραφές. Θα ήθελα να πω ότι η οδηγία έχει τεθεί σε ισχύ πρόσφατα, γι' αυτό δεν θα επανεξεταστεί στο εγγύς μέλλον. Θα ήθελα να είμαι απόλυτα σαφής. Υπάρχει πρόβλημα σε μία χώρα, στη Γερμανία, όπου μία μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία λέει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα. Και κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα σας δώσω και άλλες πληροφορίες. Και μετά από αιτήματα που λάβαμε από τη Γερμανία έγραψα στους αρμόδιους υπουργούς για να ρωτήσω ποια είναι, για να γνωρίσω τα προβλήματα, τονίζοντας ότι η οδηγία ισχύει από την πρώτη Πρώτου του τρέχοντος έτους. Και αυτό το είπα και σε μια μεγάλη εφημερίδα της Τουτγάρδη, σε μια συνέντευξή μου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στοιχεία για παραβίαση της οδηγίας από πλευράς Γερμανίας εξαιτίας αυτής της βιομηχανίας. Πρόκειται για μία βιομηχανία, μεγάλη βεβαίως. Ήρθα σε επαφή και με τους διευθύνοντες συμβούλους αυτής της μεγάλης επιχείρησης και μόνο αν δούμε ότι αυτό το ψυκτικό υγρό είναι επικίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή, κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε μέχρι τώρα, η οδηγία ισχύει. Επειδή μας ενδιαφέρει η υγεία των πολιτών και η ασφάλειά τους, λαμβάνω υπόψη όλες τις ενδείξεις και είμαι σε επαφή με τις γερμανικές αρχές. Έστειλα μία μακρά επιστολή την προηγούμενη Δευτέρα στη γερμανική κυβέρνηση Μπορώ να σας δώσω και ένα αντίγραφο, εάν το επιθυμείτε, στον πρόεδρό σας, γιατί και αμέσως σας χορηγώ αυτό το αντίγραφο. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι θέλω να ακούσω απόψεις, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει μορατόριο. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που ανέκυψαν στη Γερμανία σε αυτή τη βιομηχανία, όμως η οδηγία είναι εμπλήρη ισχύ. Όσον αφορά την πρόταση για την ηχορύπανση των οχημάτων, τη συζητήσαμε στις 5 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο και στη συνέχεια η ψήφος της Ολομελίας κατέδειξε ότι θα πρέπει να εργαστούμε επί μακρόν εάν θέλουμε να φτάσουμε σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Η Επιτροπή θέλει να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των πολιτών και γι' αυτό θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτά τα όρια εκπομπής θορύβου για τα οχήματα και τα φορτηγά. χρησιμοποιούμε τα ε, δεδομένα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, της ε, UNECE, για την προστασία των καταναλωτών. Το Κοινοβούλιο πρότεινε τροπολογίες λαμβάνοντας υπόψη την ε, ισορροπία μεταξύ εσωτερικής αγοράς και ασφάλειας των πολιτών. Κατά την άποψή μας, ορισμένες τροπολογίες αποτελούν μία βελτίωση σε σχέση με το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλες τροπολογίες που ε, αφορούν τα όρια ηχορύπανσης θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μεγάλα φορτηγά και μη ελαφρά οχήματα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πρώτη ανάγνωση. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο έτσι ώστε τάχιστα να μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτό το πλαίσιο σε δεύτερη ανάγνωση. Ο τομέας της Χαλιβουργίας επίσης μας απασχόλησε στις 12 Φεβρουαρίου το συζητήσαμε στην Ολομέλεια μετά από τη στρογγυλή τράπεζα που έλαβε χώρα στις 12 Φεβρουαρίου. Εγκρίθηκαν λοιπόν οι τελικές συστάσεις της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα προετοιμάσουν ένα σχέδιο δράσης για τη χαλιβουργία που θα εγκρίνουμε τον Ιούνιο του 2013. Στόχος είναι να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία έτσι ώστε να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη και την απασχόληση με βάση και τις κλιματικές αλλαγές. Μέσα στα πλαίσια της νέας πολιτικής υπέρ του κλίματος εν ώψη του 2020, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις τεχνολογικές και οικονομικές επιτυχίες του χαλιβουργικού τομέα και υπάρχει και ο κίνδυνος με την καταστάσεων. Εάν εγκρίνουμε ένα αυστηρό πλαίσιο μέτρων που η βιομηχανία, η χαλιβουργία δεν θα μπορέσει να τηρήσει, θα χάσουμε όχι μόνο ολόκληρα τμήματα βιομηχανίας που θα μετατοπιστούν σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά εκεί δεν υπάρχουν και αυστηροί νόμοι για την προστασία του κλίματος και έτσι θα είχαμε μία διπλή ήττα. Χάνουμε τη βιομηχανία μας και χάνουμε και μία δράση ε, καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Το σύστημα ETS, το σύστημα εμπορίας εκπομπών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά και να δούμε πώς μπορούμε να δράσουμε σε τομείς, σε τομείς υψηλής ενεργειακής ε, κατανάλωσης. Μας απασχολεί βεβαίως και η ανταγωνιστικότητα της χαλιβουργίας. Θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις έτσι ώστε να έχουμε χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα έτσι ώστε να εγκριθεί αυτό το νέο εμπορικό πλαίσιο. Υποστηρίζουμε το σχέδιο Ούλκος, δηλαδή τη χαλιβουργία χαμηλού διοξιδίου του άνθρακα και ελπίζουμε να εγκριθεί αυτό το σχέδιο τάχιστα ως προς το ΡΙΤΣ, που είναι ένας τομέας ύψης της σημασίας. Επανεξετάσαμε τον κανονισμό και η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου. Η Επιτροπή αποτίμησε και τους στόχους του ΡΙΤΣ λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές δαπάνες και το διοικητικό φόρτο των ΜΜΕ. Το ΡΙΤΣ λειτουργεί είδαμε μία μείωση του κινδύνου που απορρέει από τις ήδη καταγεγραμμένες ουσίες και το Ευρωβαρόμετρο κατέδειξε ότι το 61% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι τα χημικά προϊόντα αυτά είναι πιο ασφαλή σήμερα σε σχέση με 10 χρόνια πριν. Γι' αυτό δεν προβλέπουμε ουσιώδεις αλλαγές στο REACH Υπάρχουν όμως απαιτήσει προσαρμογής και τελειοποίησης. Θέλουμε να μειώσουμε το διοικητικό και χρηματικό φόρτο στις ΜΜΕ για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή ενέκρινε με διαδικασία επιτροπολογίας μία πρόταση τροποποίησης του κανονισμού σύμφωνα με την οποία οι ΜΜΕ θα μπορέσουν να ε, έχουν μία μείωση ε, σε σχέση με τις επιστοποιήσεις δηλαδή περνάμε από το 35% στο 95% ως προς τα ε, ποσά καταχώρησης και 25% και από 25% σε 90% σε περίπτωση πιστοποίησεων. Προσπαθούμε λοιπόν να ε, σεβαστούμε πρωτίστως το περιβάλλον. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Μιλήσατε βέβαια περισσότερο από το αρχικό δεκάλεπτο, αλλά μας αναπτύξατε θέματα που έχουν ιδίως σχέση με την ε, στρατηγική CARS 2020 Σήμερα το πρωί συζητήσαμε την έκθεση του κ. Ούλμερ που κατά τη γνώμη μου άπτεται και κάποιου πράγματος που είναι σημαντικό και που θα ήταν εναρμόνιση των φόρων. Θα, κάτι που θα ωφελήσει σημαντικά την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων που νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά θα διευκόλυνε μια κίνηση προς την ίδια κατεύθυνση. Όχι 27 ε, και σύντομα 28 διαφορετικά εθνικά συστήματα που λειτουργούν εκ παραλλήλου. Τώρα για τα υγρά ψήξεως. Είχαμε την ανακοίνωση πέρσι μιας επιχειρήσεως ότι δεν μπορεί να τηρήσει, δεν μπορεί, δεν θέλει, τέλος πάντων δεν πρόκειται να σεβαστεί την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό έχει γίνει και στη συνέντευξη τύπου. Η ερώτησή μου λοιπόν η ευρωπαϊκή βιομηχανία συμφώνησε στο 1, 2, 3, 4 YF Άρα μπορεί να το καταβαλάβει ο καθένα. Τέλο πάντων αυτό το αέριο F Εσεί παρατείνατε ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2013 θα έπρεπε να χρησιμοποιείτε αλλά ήδη κανονικά από το 2011. Από πότε λοιπόν είναι γνωστά τα προβλήματα του υγρού ψήξεως 123YF έχουν γίνει σε δοκιμασίε υπό πραγματικέ συνθήκε, όταν ο κινητήρα είναι κρύο, όταν ο κινητήρα έχει ζεσταθεί, ότι ενδέχεται το πράγμα αυτό να αναφλεγεί, ότι μπορεί να προκαλέσει, μπορεί να γίνει όξινο εφόσον οι συνθήκες έχει διερευνήσει η Κομισιόν κατά πόσο αυτό το υγρό ψύξιος έχει τις ιδιότητες αυτές υπό πραγματικές συνθήκες διότι αυτό μέχρι τώρα το έχει διερευνήσει μόνο ένας κατασκευαστής ο οποίος δεν συμμορφώνεται με, τις, ε, με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία οι υπόλοιποι τα τηρούν. Άρα αυτός ο κατασκευαστής επομένως διοχετεύει στην αγορά αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν έγκριση τύπου στην ουσία. Μπορεί η Κομισιόν να λάβει, να λάβει κάποια μέτρα για να κάνει αναξάρτητες έρευνες, δοκιμασίες και αυτά που λένε real-time test, δηλαδή με κινητήρα ζεστό το 2008 λήφθηκε δυστυχώ απόφαση κατά του δεξιού του άνθρακα ω ε, μέσου ψήξεω που δεν θα είχε τέτοια προβλήματα. Θα δώσω τώρα το λόγο στις και στους συναδέλφους μου. Έχω πρώτα στην λίστα μου Chris Davis, Σάτου Χάση, Μπόγκουσταυ Sonik, Κροστέτ. und Sophie Okuni. Habe ich Richard der EVP erhält er natürlich Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σου αυτή της εναρμόνισης της φορολογικής πολιτικής. Βέβαια δεν είναι ο σωστός συνομιλητής ο Επίτροπος Ταγιάννη. Ίσως πρέπει να φωνάξουμε κάποια στιγμή εδώ τον αρμόδιο Επίτροπο. Να αρχίσω κι εγώ λοιπόν με τα αυτοκίνητα. Από τη δική μας σκοπιά είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν όλοι οι κατασκευαστές να χρησιμοποιούν ένα προϊόν το οποίο ενδεχομένως έχει, μια, ενέχει ένα κίνδυνο και ένας και μόνος κατασκευαστής που ισχυρίζεται κιόλας ότι έχει τεχνολογική πρωτοπορία. Θεωρεί ότι αυτό είναι αδύνατον και ζητεί να εξαιρεθεί και η Κομισιόν ε, υποχωρεί απέναντί του. Βρίσκω κάπως δύσκολο να το χωνέψω αυτό. Ως νομοθέτης θα πρέπει κανείς να φανεί και σκληρός έτσι ώστε να παραμείνει μέσα στα πλαίσια μιας κοινότητας δικαίου διότι κάπου χάνουμε την αξιοπιστία μας. Βλέπω και από τις ερωτήσεις και απαντήσεις στην ιστοσελίδα της Κομισιόν ότι δεν έχει αποδειχθεί αυτή η επικινδυνότητα του προϊόντος ψήξεως και γι' αυτό παρακάλεσα τον Επίτροπο να τηρήσει αυστηρά το γράμμα της νομοθεσίας, διότι όλοι οι άλλοι που συμμορφώνονται με την νομοθεσία εν τέλει αντιμετωπίζουν συγκριτικό μειονέκτημα. Χαίρομαι και για την στατική της Κομισιόν και τη δική σας κύριε Ταγιάννη που κάνετε προσπάθεια να αποδώσετε πάλι την αξία που της αξίζει στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αλλά αυτό θα γίνει δυνατό η, ε, η Ευρώπη θα διατηρήσει την πρωτοπορία της μόνο εφόσον διατηρήσει την πρωτοπορία της η βιομηχανία. Είναι δύσκολο εδώ πρέπει να μπουν στη μέση όλες οι βιομηχανίες και η χαλιβουργία κλπ. Και είμαι βέβαιος ότι και για λόγους πολιτικής του κλίματος είναι καλύτερα να ασκήσουμε οριζόντια στάνταρτ πολιτική με φιλόδοξους στόχους ό,τι αφορά το διοξίδιο του άνθρακος, τα ε, υδάτινα λίμματα κτλ. Αλλά σε ένα πλαίσιο το οποίο να καθιστά δυνατή τη βιομηχανική παραγωγή. η Ιδεμή θα δούμε ολόκληρη διαδικασία προσθήκης αξίας να μεταναστεύει. Και αυτό δεν εξυπηρετεί βεβαίω το κλίμα και πολύ λιγότερο την απασχόληση. Αυτέ λοιπόν είναι οι βασικέ αρχέ οι οποίε με βρίσκουν σύμφωνο και έχει την υποστηρίξη τη Επιτροπή Περιβάλλοντο. Πάντω, όταν έχουν εγκριθεί κανόνε, πρέπει και να τηρούνται και σας είχα παρακαλέσει να επιμείνετε. Εκτός βέβαια και αν υπάρχουν εκτελώς, εντελώς εξαιρετικές συνθήκες που πρέπει να αποδειχθούν, αλλά μέχρι τώρα δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Chris Davis. Ε, αρχίσαμε αρκετά αργότερα αλλά, εν πάση περιπτώσει, κύριε Επίτροπε, δεν ε, μπορέσατε να θέσετε σε εφαρμογή τον ε, κοινοτικό νόμο σε σχέση με την Daimler, η οποία δεν ε, συμμορφώθηκε με αυτό το ψυκτικό υγρό. Την προηγούμενη Δευτέρα μιλήσατε για τη θέση της Επιτροπής με ένα έγγραφο ένα πολύ δυνατό έγγραφο που είναι σαν κήρυξη πολέμου κατά της Daimler. Μιλάτε για την ισχύ του νόμου που υπερέχει όλων των άλλων. Δεν επικρίνω την τρέχουσα θέση σας. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετική. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε μερικούς ότι εγώ παρακολούθησα αυτό το νόμο από όταν ε, εισήχθη το 2003. Μίλησα με τον τότε εισηγητή. Ο Επίτροπος μας μίλησε για το στόχο της νομοθεσίας. Ε, βεβαίως υπήρξαν υπεξαιρέσεις, κολυσιεργίες με συγχωρείτε, και το 2008 ε, είπαν ότι θα, θα ακολουθήσουν το δρόμο της ε, μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά το 1224 HFO δεν χρησιμοποιήθηκε Μίλησα δύο φορές με τον Επίτροπο Βερχόιγκεν για να μιλήσω για την εφαρμογή και μίλησε για το ότι έπρεπε να τεθεί σε ισχύ από την 1η Πρώτου 2011. Εσείς το παρατείνατε για δύο χρόνια. Ακόμα και τώρα αναγνωρίσουμε ότι είτε είναι ασφαλές το προϊόν, γιατί χρησιμοποιείται από την Toyota, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, ε, BMW, Land Rover και πολλές άλλες ε, εταιρείες. Μόνο η Daimler δεν το χρησιμοποιεί και λέει ότι θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιήσουμε το 134α είναι ε, ένα προϊόν το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε εκπυρσοκρότηση. Είναι έφλεκτο, με συγχωρείτε, υλικό και μπορεί να γίνει ανάφλεξη και αυτό ε, έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή η, αυτή η εταιρεία δεν δε θέλει να πληρώσει ένα επιπρόσθετο κόστος για αυτό το ε, υγρό. Μιλάμε για 20 ευρώ παραπάνω και στις ε, ερωταποκρίσεις σας αυτό ακριβώς είπατε. Ο κίνδυνος είναι ίσως και κατώτερος με άλλα τέτοια ε, ε, ψυκτικά υλικά. Όταν μιλάμε για το σύστημα κλιματισμού αυτών των οχημάτων, δηλαδή αν η Daimler έχει πρόβλημα, είναι γιατί δεν σχεδιάζει καλά τα αυτοκίνητα και το σύστημα κλιματισμού τους πολύ σαφώς είπατε σε αυτό το έγγραφο και στη δήλωσή σας, θα σας διαβάσω από το δικό σας έγγραφο, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης δεν ισχύει εάν δεν συμμορφούται το όχημα. Με το 134α η Daimler δεν τηρεί, δεν τηρεί τον ε, νόμο και γι' αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό κάτι τέτοιο για την ταξινόμηση νέων οχημάτων. Η Επιτροπή θα λάβει μέτρα κατά παρομοίων παραβιάσεων. Μιλάτε λοιπόν για τα οχήματα της Daimler από τον Ιανουάριο και αν χρησιμοποιούν το 134α τότε είναι παράνομοι και αυτό απορρέει από το έγγραφο σαφέστατα. Ο Επίτροπος είναι απόλυτα σαφής. Το ζήτημα είναι τι θα κάνετε, διότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή αυτό το νόμο. Τι θα κάνετε έτσι ώστε να συμμορφούνται τα κράτη-μέλη για να μην πολιθούν αυτά τα οχήματα. Θα εκινήσει διαδικασία επιπαραβάση αν δεν σταματήσει η πώληση αυτών των οχημάτων. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ δυνατή σας δήλωση. Σα του χάσει. Συμφωνώ με τον Chris Davis για τα κινητά ε, κλιματιστικά. Όμως υπάρχει κι άλλο ένα θέμα σχέση με τα αυτοκίνητα. Είπατε, Επίτροπε, ότι χρειάζεται περισσότερη καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία. Συμφωνώ. Και ένας τομέας ε, που χρειάζεται καινοτομία είναι ο θόρυβος. Η δήλωσή σας για το τι για αυτά ψήφισε το Κοινοβούλιο για, τα, για τις στάθμες θορύβου δυστυχώς ήταν ε, λίγο ασαφής, τουλάχιστον αυτό που άκουσα εγώ από την μετάφραση ήταν λίγο ασαφές. Ε, θα ήθελα λοιπόν σας ρωτήσω, να σας ζητήσω μάλλον να είστε αυστηρός σε ό,τι αφορά την φιλοδοξία περιστάθμισης επιπέδων θορύβου ε, στις προτάσεις να προστατεύσετε τα συμφέροντα των πολιτών και να μην μειωθούν τα όρια η, ε, η μείωση έτσι κι αλλιώς των ορίων της πρώτης Κομισιόν πέρασε με πολύ μικρή πλειοψηφία από την Ολομέλεια. Θα ήθελα να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα των πολιτών και την αρχική σας πρόταση. Ένα άλλο θέμα το οποίο σχετίζεται με κάτι που εκρεμεί είναι η... το κριτήριο βιωσιμότητας βιομάζας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, αν η αυτοκινητοβιομηχανία θα ε, προτιμούσε ε, μία προσέγγιση του τύπου cascade, δηλαδή κλάσματα της βιομάζας χρησιμοποιούνται ανάλογα με την οικονομική τους αξία και ε, χρησιμοποιούνται ε, έτσι ώστε ε, να καίγονται για παράδειγμα τα λιγότερο πολύτιμα κλάσματα της βιομάζας αυτά που είναι προς απόρριψη κατά βάση ενώ να χρησιμοποιούνται με άλλο τρόπο τα υπόλοιπα κλάσματα. Ε, τα κριτήρια επισημότητα στη χρήση της βιομάζας, όπως θα θυμάστε, δίνουν εναλλακτικές λύσεις ε, για αυτή την ε, κλασματική χρήση. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος συντονιστής τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τον Επίτροπο Ταγιάννη. Είμαι πολύ ικανοποιημένο από τις δηλώσεις του σε σχέση με τα ψυκτικά υγρά στα οχήματα. Δεν έγινε παράταση και τώρα όπως είπατε όλοι θα πρέπει να συμμορφωθούν με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ως προς την ηχορύπανση από τα οχήματα θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα επαχθές και δαπανηρό το σύστημα που ορίζει η Επιτροπή. Θα προτιμούσα το αρχικό κείμενο. Σε σχέση με το πρόγραμμα δράσης για την χαλιβουργία είναι κάτι το απόλυτα αναγκαίο. Εμείς στην Ιταλία, η Ιταλία καταβάλει 400% περισσότερο για ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με την ίδια επιχείρηση που παράγει χάλιβα ε, και εδώ μιλώ για τις ΗΠΑ, όχι για την Αμερική γενικότερα. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι η Αμερική είναι ο τρίτος κόσμος. Γι' αυτό υπάρχει κίνδυνος μετεγκατάστασης αυτών των επιχειρήσεων. Ως ε, προς τις πληροφορίες που μας δώσατε μέσα στα πλαίσια της επιτροπολογίας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ. Ε, πολύ καλό αυτό το βήμα. Ο Επίτροπος να απαντήσει στον πρώτο γύρο. Εντάχει. Και θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Θα προσπαθήσω εντάχει. Ως προς το θέμα του ψυκτικού υγρού. Δεν μπορώ να σας διαβάσω την επιστολή που απέστειλα στη γερμανική κυβέρνηση, γιατί είναι χρονοβόρο. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οδηγία έχει τεθεί ισχύ από την 1η Πρώτου του 2013 και θα τηρηθεί. Εάν ε, λάβω στοιχεία για παραβίαση της οδηγίας, από οποιοδήποτε κράτος μέλος θα ανοίξει η ε, προσήκουσα διαδικασία. Λάβαμε από την γερμανική κυβέρνηση ένα αίτημα και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες σύμφωνα με τις οποίες η Daimler, στη Daimler μάλλον, ε, ανοιχνεύτηκαν στοιχεία επικινδυνότητας του ψυκτικού υγρού αυτού. Με βάση αυτή την κοινοποίηση ενδεχομένου κινδύνου, είναι καθήκον μου να δράσω, ακόμα και αν πρόκειται για εξαίρεση, γιατί οι άλλες, τα άλλα στοιχεία καταδεικνύουν το αντίθετο. Δεν μπορώ όμως να μην ανησυχήσω. Τις προάλλες έγραψα δύο επίστολες στην, ε, στον Υπουργό και στον ε, ε Καγκελάριο Ρέσλετ και τον αναπληρωτή Καγκελάριο Ρέσλερ για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Και ζήτησα στοιχεία. Και επανέλαβα ότι η οδηγία βρίσκεται ισχύ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ εμπλεκομένων βιομηχανιών γιατί έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Γι' αυτό και εφήγει αυτό το θέμα ουσίας. Στην επιστολή ζητώ ακριβείς πληροφορίες από τη γερμανική κυβέρνηση για ενδειχόμενα στοιχεία ως προς την επικινδυνότητα του ψυκτικού υγρού. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν ισχύει η οδηγία. Ε, περιμένω την απάντηση από τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Καγκελάριο. Εφόσον λοιπόν είχαμε μία κοινοποίηση για την επικινδυνότητα, θεωρώ ότι πρέπει να ζητήσω περαιτέρω πληροφορίες και να τις αποτιμήσω. Αναμένω απάντηση από την γερμανική κυβέρνηση και έχετε στη διάθεσή σας τις επιστολές. Ως προς το ε, θέμα του, της συγχωρήπανσης στα οχήματα, Ίσως η κυρία Χάση δεν άκουσε σαφώς τη θέση μου. Επαναλαμβάνω αυτά που προείπα. Αργά και καθαρά, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Αξιολογούμε όλες τις τροπολογίες ε, που έχουν προταθεί από το Κοινοβούλιο. Όπως ανακύπτει και από την παρέμβαση του κύριου Ρώση, δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση ε, ούτε από την ΕΜΒΗ ούτε από το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό θα ήθελα να επιτύχουμε κάποια εξισορρόπηση μεταξύ ενιαίας αγοράς προστασίας του περιβάλλοντος και προστασίας της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών και παράλληλα να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός και στα τρία αυτά μέτωπα. Προσωπικά, ορισμένες τροπολογίες ε, αποτελούν βελτίωση του αρχικού κειμένου της Επιτροπής. Αναφέρομαι στην ε, προσαρμογή του κειμένου στα στοιχεία της ΟΝΕΤΣΕ, δηλαδή της ε, Οικονομικής Επιτροπής ε, των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη. Υπάρχει και, και τα όρια ηχορύπανσης για τα λεωφορεία, για τα φορτηγά και για τα αυτοκίνητα σπορ. Θα πρέπει λοιπόν να αποτιμήσουμε την, ε, τις επιπτώσεις και για αυτές τις ε, κατηγορίες. Εμείς ως ε, μεσολαβητές θέλουμε να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό αν και είναι δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Όπως σας είπα, ορισμένες τροπολογίες κινούνται προς τη μία κατεύθυνση, ενώ άλλες προς την αντίθετη όπως ανακύπτει και από τη συζήτηση, υπάρχει διχογνωμία. Γιατί η δική σας θέση δεν είναι η ίδια με του κυρίου Ρώση. γιατί και εκείνος αναφέρθηκε στο θέμα της αυτοκινητοβιομηχανίας ως προς τη χαλιβουργία και το κόστος της ενέργειας είναι ένα θέμα που με απασχόλησε και σήμερα γιατί ζήτησα από τον πρώην Επίτροπο Νταβινιών, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος Επίτροπος που μπορούσε να ασχοληθεί με αυτή την αναδιάρθρωση της χαλιβουργίας. Ασχοληθήκαμε και με το ενεργειακό κόστος. Θα ξαναμιλήσω με τον Επίτροπο Έτιγκερ Αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί που θα λάβουμε υπόψη και για το πρόγραμμα δράσης που θα παρουσιάσω στο Διευθυντήριο μέχρι τα τέλη Μαΐου. Ευχαριστώ για την απάντηση των ερωτήσεων. Αυτά για τα κλιματιστικά μηχανήματα 123YF το οποίο έχει, αυτό είχα ρωτήσει, αν το έχει εξετάσει η Κομισιόν με συνθήκες πραγματικές, δηλαδή με θερμό κινητήρα. Βεβαίως, η θέση μας είναι ότι για αυτά τα ψυκτικά υγρά δεν υπάρχουν κίνδυνοι ψηλότεροι από οποιονδήποτε άλλο. Αυτά δείχνουν οι δοκιμέν μας. Εάν όμως μία κυβέρνηση, ένα κράτος μέλος μου κοινοποιήσει ένα θέμα, θα πρέπει να ασχοληθώ. Αυτό όμως ε, δεν σημαίνει ότι εφαρμόζω ε, εξαιρέσεις ή κάποια εξαίρεση. Ζητώ περισσότερες πληροφορίες από τη γερμανική κυβέρνηση. Ωραία, σαφής απάντηση και σαφή ερώτηση. Είναι καλό που έχουμε την πληροφορία αυτή. Τώρα, Σόνικ, Γκροστέτ, Περίλο, Κονί και Γκερμπράντι. Σόνικ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Ταγιάννη. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Μπαρόζο, πριν από μερικούς μήνες μας είπε ότι η θέση Κομισιόν για το σχιστολιθικό αέριο και ε, ε, θα καθοριστεί από τέσσερις επιτρόπους μαζί, συναρμόδιους, περιβάλλοντος, ε, οικονομίας, βιομηχανίας. και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς εμπλέκεστε σε αυτή τη μελέτη θα ήθελα να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία στη θέση τη Κομισιόν για αυτό το θέμα του σχιστολιτικού αερίου. Ευχαριστώ κύριε Γκροστέτ. Μια παρατήρηση και μια ερώτηση. Σε ό,τι αφορά το, τα ψυχτικά υγρά, ε, είσαστε πολύ ρητός και κατηγορηματικός. Ε, μπράβο γι' αυτό. Θέλουμε όμως να το κάνετε μέχρι το τέλος αυτό, να κρατήσετε την διαστάση. Γιατί η γερμανική κυβέρνηση μπορεί να καθυστερήσει εβδομάδε να σα απαντήσει. Εν τω μεταξύ, εμείς βρισκόμαστε σε ενώπιον μιας κατάστασης αθέμητου ανταγωνισμού μεταξύ ενός κατασκευαστή απομονωμένου στην Ευρώπη και όλων των υπόλοιπων που έχουν κάνει τις προσπάθειες να εφαρμόσουν την οδηγία και που μας λένε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό το ε, ψυχτικό υγρό. Συνεπώς, ε, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, παρακολουθούμε πολύ στενά το τι θα κάνετε. Δεν πρόκειται να μας τη φέρει μια κυβέρνηση που ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα ε, τις ερωτήσεις αυτές ε, για να, τα ερωτήματα αυτά για να καθυστερήσει. Το θέμα δεν αφορά πλέον μόνο την αυτοκινητοβιομηχανία, ε, αλλά και, μάλλον το άλλο θέμα αφορά τη φαρμακοβιομηχανία. Ε, τον Οκτώβριο 2012 δημοσιεύσατε ένα κείμενο για το μέλλον της ε, φαρμακοβιομηχανίας και προτείνατε να ξεκινήσει ένα στρατηγικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των φαρμακευτικών προϊόντων. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε πού βρίσκεται η, η του θέματος αυτή τη στιγμή και τι θα λέγατε στο, στην, για την πρόταση να δημιουργηθεί μια ειδική ομάδα εργασίας στην οποία θα συμμετείχαν και μέλη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερα την αποφασιστικότητα του Αντιπροέδρου Ταγιάννη ε, ως προς την εφαρμογή της οδηγίας που έχει τεθεί σε ισχύ από την πρώτη πρώτου του τρέχοντος έτους. Εκτιμώ και με τη σαφήνεια γιατί με την οποία μίλησε είπε δεν υπάρχει μορατόριο, δεν υπάρχει αναπομπή, δεν υπάρχει παράταση. Πολύ σωστά έλαβε υπόψη και μία μεμονωμένη περίπτωση και δεν υποχώρησε. Θα έπρεπε να υπάρξουν κυρώσεις για αυτούς που έθεσαν σε, σε χρήση αυτό το προϊόν. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι στεναρή η στάση μας για να δείξουμε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, όπως είπε και ο Επίτροπος με μεγάλη σαφήνεια. Ευχαριστώ. Η Σοφία Κονή. Πολλά ελέγχθησαν, Πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που όλο ένα και αλλάζει. Από το 8 και μετά είδαμε ότι έχουμε χάσει τρία εκατομμύρια ε, θέσεων απασχόλησης και ε, έχουμε πρότυπα ανταγωνιστικότητας που σημαίνουν μεγάλες ε, αλλαγές. Οι αναδιόμενες οικονομίες αποτελούν βασικούς παράγοντες και κινητήριο δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας. Εμείς θα πρέπει να υποστηρίξουμε την πράσινη οικονομία, την πράσινη βιομηχανία και την πράσινη ανάπτυξη. Έτσι θα μπορέσουμε να, βρούμε, ε, να ξαναβρούμε την οδό της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους οικονομικούς μοχλούς ε, για την έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη με βάση την περιφερειακή πολιτική ή την έκκληση για σχέδια. Αυτό θα πρέπει να δει και το ΕΤΠΑ, γιατί μιλάμε για ένα 40, 65 με των επιχειρήσεων που ε, εμπλέκονται σε θέματα ανταγωνισμού. Αυτό είναι ένα πλαίσιο πολύ δύσκολο για τις επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε πλήρη απασχόληση και δυστυχώς η, εικόνα της Ευρώπης φθήνει, διότι δεν έχουμε απλουστεύσει και τη γραφειοκρατία μας. Ας απλουστεύσουμε, ας επιταχύνουμε αυτές τις ε, διαδικασίες με λιγότερη γραφειοκρατία, διότι σε μια κατάσταση κρίσης θα πρέπει να λάβουμε και έκτακτα μέτρα. Διαφορετικά θα καταρρεύσουν οι βιομηχανίες μας θα πρέπει να πλουστεύσουμε αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες τη στιγμή που ξέρουμε ότι υπάρχουν τα χρηματοοικονομικά μέσα. Κέρμπραντι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ταγιάννη και τον Ενθαρρύνω να προσέρχεται ενώπιον μας συχνότερα διότι η ανταγωνιστικότητα της ε, βιομηχανίας όλο και περισσότερο αποφασι... κρίνεται μάλλον από το επίπεδο βιώσιμης παραγωγής της ε, βιομηχανίας. Ο κ. Ποτότσνικ χθε σε μια ομιλία του εξήγησε ότι αυξήθηκαν οι τιμές των ε, πρώτων υλών πάνω από 300% στην τελευταία δεκαετία και ότι σε προηγούμενες δεκαετίες η βασική, ο βασικός στόχος ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Τώρα όμως η παραγωγικότητα των πόρων, δηλαδή των πρώτων υλών, ίσως είναι το κύριο που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Και η ερώτησή μου αναφέρεται σε αυτό, resource efficiency. Εσείς είστε ιδιαίτερα δραστήριο, δραστήριο μέλος του resource efficiency panel. Ωστόσο, προτάσεις οι οποίες θα έπρεπε να προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστερούν είτε μιλούμε για το eco-design, είτε για ελάχιστα ποσοστά ανακύκλωσης. το Phosphorus Green Paper και άλλα. Δεν φτάνουν εν τέλει προτάσεις σας ούτε στο Συμβούλιο ούτε στο Κοινοβούλιο. Και επειδή είστε από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές, ελπίζω, της ε, ε, αποδοτικής χρήσης των πόρων, διερωτώ με εάν θα αγωνιστείτε να προχωρήσουν οι, προ... προτάσεις σας αυτές πολύ ταχύτερα και να προωθηθούν δηλαδή στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Χερμπράντι. Έχουμε φτάσει στο τέλος ε, του δευτέρου γύρου των ερωτήσεων και θα δώσω το λόγο τώρα στον ε, Επίτροπο για να μπορέσει να απαντήσει. Θα απαντήσω στα γαλλικά στην κυρία Κροστέτ ε, για να είμαι σαφής. Σε ό,τι αφορά την επιστολή που έστειλα στην γερμανική κυβέρνηση, Λέω εκεί σαφώς ότι η οδηγία έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013. Δεν δίδεται καμία πρόσθετη προθεσμία, καμία παράταση. Η οδηγία θα πρέπει να τύχει σεβασμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι η Γενική Διεύθυνση, δεν ξέρω ποιου Γερμανικού Υπουργείου, ανέφερε προβλήματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των επιβατών, είμαι υποχρεωμένος να ρωτήσω ποια είναι τα δεδομένα. Τους ζήτησα να μου δώσουν πληροφορίες. Δεν έδωσα, δεν έδωσα καμία παράταση και δεν δείχνω καμία δυναμία. Αν εσείς πάρετε μια επιστολή που αναφέρει προβλήματα υγείας, ε, δεν πρέπει να αντιδράσει. Ακόμα και αν υπάρχουν κείμενα τη Κομισιόν που αποδεικνύουν το αντίθετο. Εγώ είμαι υποχρεωμένο να ζητήσω, να ρωτήσω την γερμανική κυβέρνηση τι συμβαίνει. Δώστε μου περισσότερες πληροφορίες. Όμως αυτό δεν αλλάζει την απόφαση που ανακοίνωσα εδώ πριν από μερικού μήνε. Και το είπα και σε συνέντευξή μου στην Stuttgart, ε, σε μια εφημερίδα της Stuttgart, δεν θυμάμαι τώρα προχτέ. Ή πριν από δύο μέρε, σε πάση περιπτώσει, προχτέ. Ότι η πριν απο δυο μερε σε παση προχτες οτι η οδηγια ισχυει Και αν μου αναφερθεί ότι στην Γερμανία κυκλοφορούν αυτοκίνητα που δεν ε, σέβονται τους κανόνες και η Γερμανία έχει ε, εγκρίνει την θέση τους σε, ε, στην αγορά, ε, θα ε, ξεκινήσουμε διαδικασία επί παραβάση. Το λέω στα γαλλικά και στα ιταλικά και αν θέλετε και στα ισπανικά, κυρία Σέντερ. Νομίζω όμως ότι είναι σαφές. Η οδηγία είναι σε ισχύ. Ε, παντώ και στην κυρία Οκόνη. Στα γαλλικά συμφωνώ μαζί σας. Ε, ε, προσπάθησα να το αποδείξω στο REACH, μειώσαμε, έχουμε μειώσει με την απόφαση επιτροπολογίας ε, την ε, φορολογική, φορολογικό βάρος, δηλαδή ε, το, τα τέλη πληρώνουν οικονομικές επιχείρησεις για την καταγραφή, για την καταχώρηση και επιτρέψαμε την χρήση όλων των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληροφόρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να γλιτώσουν, να εξοικονομήσουν πόρους. Σε ό,τι αφορά την ε, ε, γραφειοκρατική απλοποίηση αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ορίζον 2020, κόσμε, ήδη όταν ήμουν επιτροπός μεταφορών, το είχα κάνει και στο Σιωτεφρά το Μαρκο Έχουμε προσπαθήσει να απλοποιήσουμε την συμμετοχή σε όλες τις ε, προσκλήσεις εκδήλωση ενδιαφέροντος ε, ε, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, να απορροφηθούν τα ποσά τα οποία έχει δεσμεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. η απλοποίηση της ε, η γραφειοκρατική απλοποίηση είναι πλέον ευθύνη του Προέδρου της ε, Επιτροπής αλλά προσπαθούμε, εγώ προσπαθώ να ε, διευκολύνω, να απλοποιήσω τις διαδικασίες σε όλους τους τομείς. Είναι, έχω δεσμευτεί ως προς αυτό. Απαντώ και στο ερώτημα και την έκθεση του κύριου Γκέρμπραντι να προσέρχομαι συχνότερα. Το κάνω με μεγάλη ευχαρίστηση. Ξέρετε ότι ήμουνα Ευρωβουλευτής για 15 χρόνια. Γι' αυτό ε, αποτελεί μεγάλη χαρά για μένα να προσέρχομαι και να συζητώ μαζί σας με σας τους πρώην συναδέλφους. Συνεργάζομαι με τέσσερις, τέσσερις επιτροπές είτε για θέματα eco-design, είτε για αποδοτικότητα των, ως προς τη χρήση των πόρων. Θα ζητήσω να επιταχύνουμε τη διαδικασία και ως προς τις δικές μου αρμοδιότητες για το θέμα eco-design Ξέρω ότι η διαδικασία έγκρισης ήταν χρονοβόρα και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να έχουμε κοινά πρότυπα για την ε, κατηγορία προϊόντων υπορρύθμιση λαμβάνοντας υπόψη τη θέση των εμπλεκομένων φορέων. Όσον αφορά την οδηγία Eco Design, νομίζω ότι Οι τρεις νομοθετικές πράξεις ε, θα εγκριθούν φέτος και η περίοδος εργασίας 12-14 σχετίζεται με την ε, θερμική μόνωση, ε, παράθυρα και άλλα μονοτικά υλικά. Και αυτό είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα. Όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Σόνικ, για ενεργειακά θέματα, τα οποία συζήτησα με τον Επίτροπο Έτιγκερ. Συνεργαζόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε βιομηχανική πολιτική αν δεν έχουμε και ενεργειακή. Δεν έχω συγκεκριμένες ε, πληροφορίες επί του θέματος, αλλά μόλις τις ε, λάβω θα σας τις κοινοποιήσω. Θα αναφερθώ λοιπόν στον υπεύθυνο για να ζητήσω διασαφήσεις. Υπήρχε και ένα άλλο ζήτημα σε σχέση με, τα, ε, με τον φαρμακευτικό ε, κόσμο. Υπάρχει μία ομάδα που εργάζεται για τη διαφάνεια των τιμών. Εστιάζουμε την ε, προσοχή μας στην Αφρική και ως προς τη συμμετοχή των Ευρωβουλευτών δεν έχω πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς αποφασίζετε για τη συμμετοχή ε, ευρωβουλευτών στην εργασία της Επιτροπής, αλλά με μεγάλη χαρά να σας δεχτώ να με βοηθήσετε να βρούμε τις κατάλληλες, τις καταλληλότερες ε, λύσεις για όλους. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, αν υπάρχουν άλλα θέματα να σας ακούσω με ενδιαφέρον. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν μόνο προκλήσεις και δυνατότητες λύσεων. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έρχεστε σε ένα σώμα 744 εκλεγμένων εκπροσώπων που εργάζονται σκληρά προς το συμφέρον και την προστασία των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Βεβαίω και πολλά, για πολλά θέματα τα οποία εμπίπτουν στο δικό σα χαρτοφυλάκιο. Στην εισαγωγή σα εξηγήσατε ότι αντιμετωπίζουμε όντω μεγάλε προκλήσει και σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα. Εγώ δεν μιλώ για green economy, είναι δύσκολο να τα εξηγήσει κανεί αυτά στον κόσμο. Μιλώ για την ανάγκη διαμόρφωσης βιώσιμης οικονομίας προς τις τρεις κατευθύνσεις. Είστε πάντοτε ευπρόσδετος εδώ. Σας ευχαριστώ που προσήλθατε και μας επιτρέψατε έτσι να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Ja, jetzt geht es weiter nach dem... Προχωρούμε τώρα μετά την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ταγιάννη. Προχωρούμε τώρα στο επόμενο θέμα στον εισηγητή κύριο Μπαρτολόση βιοοικονομία για την Ευρώπη. Ο κύριος Πάολο Μπαρτολότσι είναι εισηγητής της εκθέσεως ε, ιδίας πρωτοβουλία, λαμβάνει αμέσω τον λόγο για να εξηγήσει τα της εκθέσεω. Περιμένουμε λίγη ώρα ώστε να μπορέσουν να αποχωρήσουν όσοι δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται να συμμετάσχουν στη συζήτηση, για να μπορέσει ο συνάδελφό μας να κάνει τη δουλειά του μέσα σε περιβάλλον ευπρεπέ. Έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ένα χρόνο, εδώ και ένα χρόνο η Επιτροπή ενέκρινε ε, μία έκθεση μιλώντας για την καινοτομία, ε, για μία βιώσιμη ανάπτυξη έτσι ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε σε ένα βιωσιμότερο πλαίσιο χρήσης των πόρων με βάση τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα 40 χρόνια. Η αύξηση του παγκοσμίου πληθυσμού και η μεγαλύτερη ζήτηση ενέργειας και τροφίμων καθώς και η σπάνιδα ε, παγκοσμίων φυσικών ε, αποθεμάτων μας δείχνουν ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και γι' αυτό η βιοοικονομία αποτελεί μία πραγματική ε, ευκαιρία. Μιλάμε για ένα οικονομικό σύστημα που αφορά τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας για να ανταποκριθούμε στον ενεργειακό και βιομηχανικό τομέα με βάση βιοπροϊόντα για την γενικότερη βιωσιμότητα. Πρόκειται για μία οικονομία η οποία θα οδηγήσει σε μια ευφύ ανάπτυξη και θα δώσει απαντήσεις στις πρόσφατες ε, προκλήσεις. Μεγαλύτερη βιωσιμότητα αλλά και στον αγροτικό τομέα. Ε, λιγότερες εκπομπές ε, θερμοκηπίου και μεγαλύτερη κερδοφορία της αγοράς η στρατηγική για τη βιοοικονομία α, ίσως μας βοηθήσει έτσι ώστε να μην εξαρτώμεθα από ορυκτά καύσιμα και να προωθήσουμε την ε, οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Πρόκειται για έναν κύκλο εργασιών 2 δις και αφορά 22 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ξεκινώντας από αυτές τις ε, υποτιμι... Ε, αποτιμήσεις, με συγχωρείτε, ε, δέχτηκα με μεγάλη χαρά την ανακοίνωση της Επιτροπής. Πρόκειται για μία διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος και πρόκειται και για ένα πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή της ίδιας της στρατηγικής. Η υποστήριξη αυτού του τομέα αποτελεί επένδυση για το μέλλον και η Ευρώπη μπορεί να κατέχει ηγετικό ρόλο. Θα πρέπει να εξεύρουμε τις κατάλληλες υποδομές για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα πρέπει να είμαστε πλέον καινοτόμοι διότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αποτελέσματα με βάση ερευνητικές διεργασίες. Χρειάζονται λοιπόν οι βάσεις ενός κανονιστικού ρυθμιστικού πλαισίου με διεπιστημονική και πολυεπίπεδη προσέγγιση όλων των πολιτικών που εντάσσονται στην βιοοικονομία. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να έχουμε μία πολυεπίπεδη προσέγγιση με ανταλλαγή απόψεων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών έτσι ώστε να υπάρχουν συνέργειες και κοινέ στρατηγικές στον τομέα της ανάπτυξης. Επίσης, θα πρέπει να συμμετέχουν πολίτες και τελικοί χρήστες γιατί σχετίζονται άμεσα με αυτά τα ε, προϊόντα. Όπως ορίζει και το πλαίσιο δράσης της Επιτροπής, θα πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα μέσα υποστήριξης των επενδύσεων στο βιομηχανικό τομέα. Μείωση της γραφειοκρατίας, αύξηση της επιχειρηματικότητας, εγγύηση των δημοσίων διαγωνισμών έτσι ώστε να προωθήσουμε μία ισχυρή αγορά βιοοικονομίας. Με βάση λοιπόν τις βιομηχανικές υποδομές, τη, τα βιοδηληστήρια και τη συνέργεια μεταξύ τοπικού και βιομηχανικού τομέα, με τη χρήση επίσης βιομάζας θα μπορέσουμε να κάνουμε βασικά βήματα προς τα εμπρός για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και να βοηθήσουμε τις αγροτικές περιοχές με την ανάκτηση των γεών που δεν καλλιεργούνται. Υποστηρίζουμε και τις εταιρικέ συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να μπορέσουν να παρέμβουν. Χρειάζεται μια τέτοια σύμπραξη, ιδιαίτερα στον τομέα των, βιο... Ε, των βιομηχανιών, ε, βιολογικού χαρακτήρα, υποστηρίζοντας νέα σχέδια, προωθώντας νέα προϊόντα, τα οποία ε, θα δημιουργήσουν μία νέα αλυσίδα αξιών και προωθώντας καινοτόμα σχέδια αριστείας. Για αυτούς τους λόγους ε, υπέβαλα αυτό το κείμενο που τονίζει τη σημασία της συντονιστικής αυτής διεργασίας, πιστεύοντας ότι δεν θα φυσθούμε μέσον έτσι ώστε να επιτελέσουμε αυτή τη μεγάλη πρόοδο ανάπτυξης και ε, προώθησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ευχαριστώ. Θα ακολουθήσουν τώρα οι σκιώδεις εισηγητές. Παρακαλώ να περιοριστεί κάθε σκιώδης εισηγητής σε ένα δίλεπτο, ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά και να έχει ο εισηγητής να, την δυνατότητα να απαντήσει σε ενδεχόμενες ερωτήσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, λέει η κυρία Μέρκης. Γνωρίζουμε ότι τα ορυκτά καύσιμα γίνονται όλο πιο σπάνια. Θα πρέπει να βρούμε μια, έναν τρόπο να τα αντικαταστήσουμε και η βιοοικονομία μας ε, δίνει μια ευκαιρία. Ε, αλλά όχι μόνο ενεργειακά και σε επίπεδο ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης. Ταυτόχρονα πρέπει να απαντήσουμε και σε ε, σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις. Ας είμαστε όμως προσεκτικοί μπορεί να συνεχίσουμε να παράγουμε και να καταναλώνουμε ε, ε, αλλά ε, δεν θα ήταν καλό αυτό να γίνει χωρίς αλλαγή στην συμπεριφορά μας διότι έτσι θα ήταν σαν να αντικαθιστούμε κάτι με κάτι ισοδύναμο γιατί ακόμα και τα βιοκαύσιμα ή βιοοικονομία χρησιμοποιεί πόρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα αλλού ενδεχομένως. Συνεπώς η βιοοικονομία θα πρέπει να υλοποιηθεί σωστά με σωστές ευρωπαϊκές ε, πολιτικές, κριτήρια βιωσιμότητας, ε, ε, θεμητό ανταγωνισμό και μακροχρόνιο σχεδιασμό. Θα πρέπει να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των βιοηλικών. Θα πρέπει επίσης να πάρουμε υπόψη κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. να κάνουμε διάκριση ε, μάλλον να έχουμε ξεκάθαρους στόχους ε, και τα προγράμματα αυτά θα, για να είναι ρεαλιστικά θα πρέπει να ε, μειώσουμε την γραφειοκρατία. Και οι μονοπευθυντικές στηρίδες είναι πολύ σημαντικό εργαλείο έτσι ώστε όλα να γίνονται σε ένα σημείο. Αυτό θα είναι πολύ καλό, ιδιαίτερα για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Να συγχαρώ τον εισηγητή για την πολύ καθαρή του έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Γκερμπράντι. Στα Ολλανδικά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προ είχα πάει στο Πανεπιστήμιο του Χρόνιγκεν και εντυπωσιάστηκα πολύ από τις διάφορες δυνατότητες που μου έδειξαν για τη χρήση της βιομάζας ή πια μπύρα σε ένα πλαστικό ποτήρι το οποίο είχαν φτιάξει από βιομάζα και το πέταξα μετά διότι ε, ήταν βιοαποδομήσιμο επειδή μπορούσε, ήταν φτιαγμένο από βιομάζα. Το ίδιο για ε, γλάστρες που είναι ένα είδος πλαστικού το οποίο όμως είναι φτιαγμένο από βιομάζα και μάλιστα το φυτό ε, αντλεί και συστατικά και από την ίδια τη γλάστρα. Αυτά προδεκαετίας. Από τότε έχουμε δει πολλέ καινοτόμε επιχειρήσεις, μικρές βεβαίω, αλλά και μεγάλη κλίμακα που έχουν προωθήσει φιλόδοξα σχέδια και εξετάζουν, εξετάζουν μια ε, οικονομία με βιολογική βάση. Διαβάζοντας ωστόσο την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπω να μου αυτό που βλέπω να λείπει δηλαδή είναι η υπόσχεση για το μέλλον καθώς και κάποιος επίγον χαρακτήρας. Και βρίσκω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο κρίμα. Βεβαίω και υπάρχουν πολλά καλά στο έγγραφο, αλλά βλέπω να λείπει ακριβώς αυτό. Μια αίσθηση επίγοντος, ότι δηλαδή πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτερα, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα κριτήρια καθώς και στην cascading της, στο cascading της ε, ε, βιομάζας, δηλαδή τη διαδοχική χρήση των ε, διαφόρων ειδών βιομάζας για διαφορετικούς σκοπούς. Την κλιμακωτή χρήση της βιομάζας. Έχω την πρόθεση πάντως για τα κριτήρια βιωσιμότητας να καταθέσω τροπολογίες. Ευχαριστώ τον κύριο Μπαρτολότσι για την θαυμάσια εκθεσή του. Επί ορισμένων παραγράφων είχα σκοπό να υποβάλω τροπολογίες, αλλά ήδη βρίσκω αυτά που ήθελα στην έκθεσή του. Βεβαίω, θεωρώ ότι η έκθεσή του είναι σημαντική συμβολή προς την κατεύθυνση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής. Ευχαριστώ Γιάννη. Ο κύριο Μπασάχερτ. Σαν να μιλούν όλα Ολλανδοί με Ολλανδούς. Ίσως επειδή όταν συζητούμε την βιοοικονομία ε, ε, ε, υπάρχουν πολλές Ολλανδικές εταιρείες οπότε μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ε, πάντως μας δίνεται η ευκαιρία να ξεφορτωθούμε αυτή την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιώντας βιομάζα. Ε, οπότε ε, υπάρχει μια, και μια οικολογική διάσταση αλλά για να σταθούμε στην, στον, στην ανακοίνωση της Κομισιόν και στην έκθεση ε, και στον εισηγητή ε, και στα δύο κείμενα αναφέρεται ότι η ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη, αλλά ο τίτλος λέει βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεπώς το ερώτημα είναι θα χρησιμοποιήσουμε τη βιομάζα με βιώσιμο τρόπο. Και ένα από τα προβλήματα της βιομάζας είναι ότι θα, στο μέλλον, θα γίνει πιο σπάνια, πιο σπάνιος πόρος. Ήδη είναι, θα γίνει ακόμα περισσότερο, αλλά στην έκθεση δεν αναφέρεται η βιώσιμη ανάπτυξη, διότι αν όλοι μας τρέξουμε και βιαστούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βιομάζα και δεν το κάνουμε με βιώσιμο τρόπο, δεν το κάνουμε με όρια, με, δεν το κάνουμε με σεβασμό στα όρια που μας δίνει η φύση, τότε θα αποτύχουμε. Και η κυρία Μάρκη και ο κύριος Γερμπράντη μίλησαν για την κλιμακωτή χρήση τη βιομάζα. Είναι πολύ κρίσιμο σημείο. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ε, η, το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ποσότητα βιομάζα χρησιμοποιείται ε, στον ενεργειακό τομέα. Αυτό είναι προβληματικό. Θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Δεν θέλουμε να δώσουμε κίνητρα σε μη αποδοτική ή λίγο αποδοτική χρήση της βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας. Αυτό καταστρέφει. 4 και 53 έχω φτάσει. 4 και 53 Περνάει ο χρόνος πολύ γρήγορα. Ε, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει επίσης να αναχρησιμοποιούμε ε, τα υπολείμματα της βιομάζας από την, που προκύπτουν από την πρωτογενή της χρήση. Λοιπόν, αν χρησιμοποιήσουμε τη βιομάζα βιώσιμα, ναι, μπορούμε να βγούμε από τον φαύλο κύκλο της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η βιομάζα με τον, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκεί που δίνει τη μεγαλύτερη δυνατή προσθέμενη αξία. Διαπιστώνω ότι συνάδελφοι από την Ολλανδία έχουν ήδη καταναλώσει 15 λεπτά χρόνο. Η κυρία Ρόσμπαχ που εκπροσωπεί σήμερα όλους τους υπολείπους της ECR, μόνη της εδώ στο Μετερίζι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, βέβαια εκπροσωπώ την κυρία Ρούσκη, αλλά μετά έχω και δικά μου να πω. Η κυρία Ρούσκη μου είπε να πω ότι η, χαιρετίζει τη διεύρυνση του σχεδίου δράσεως από πλευράς του συντονιστού και το πρόγραμμα της εκπαίδευσης για τη βιομάζα πρέπει να γίνει και στο επίπεδο των χωρών μελών, των χωρών δηλαδή, αλλά και των περιφερειών και των τοπικών συνθήκων, ώστε να είναι εγγύς του πολίτου. Επίσης, ζητούν, ζητεί η συναδελφός μου υποστήριξη των μέσων για την προστασία της ε, υφιστάμενης παραγωγής και για κοινοπραξίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο ιδιωτικός τομέας να ε, προσεγγίσει τον δημόσιο τομέα υποβάλλοντάς του ιδέες. Εμείς χαιρόμαστε που ο εισηγητής εγκύπτει στο θέμα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. Και μένα με χαροποιεί ιδιαίτερος προσωπικά το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια καλύτερη αξιοποίησης των απορριμμάτων και αποβλήτων. Οι δικέ μου τώρα παρατηρήσει. Χαίρομαι ιδιαίτερω για το γεγονό ότι η Κομισιόν επιλαμβάνεται του θέματο με τόσο σοβαρό τρόπο ώστε πέντε συνολικά γενικέ διευθύνσει εγκύπτουν στο θέμα. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι η Ευρώπη αλλά και ο υπόλοιπο κόσμο αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερη σπάνιδα των πόρων και αυτό θα ενταθεί στο μέλλον. Γι' αυτό και πρέπει να γίνει προσπάθεια πολύ καλύτερης χρήσης των πόρων και σεβασμού τους. Αυτό που βλέπω επίσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. Είναι πολύ σημαντική. Βέβαια πρέπει αυτό να γίνει κυρίως σε βιολογική βάση. Ο συνάδελφος Χερμπραντή είπε ορισμένα ενδιαφέροντα πράγματα και η Σουηδία όμως έχει μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τις βιολογικές καινοτομίες. Ευχαριστώ κυρία Ρόσπαχ, η κυρία Άντερσον από την Ενωτική Αριστερά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή καταρχήν για τη δουλειά που έχει κάνει. Έχω όμως κάποιες επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του και την προσέγγιση της Κομισιόν για τη βιοοικονομία. Πιστεύω ότι θα, θα πρέπει να μελετούμε καθαρέ εναλλακτικέ λύσει αλλά όχι οποιαδήποτε εναλλακτική λύση, ούτε να αναζητούμε μία λύση για όλα τα προβλήματα. Πριν ενθαρρύνουμε του ε, πολίτε και του παραγωγού ε, να αγκαλιάσουν την παραγωγή τροφίμων με βιοενέργεια, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ε, θα είναι ασφαλή τα τρόφιμα. Η αντιμετώπιση αύξηση του προπολογισμού και τη αύξηση τη ζήτησης τροφίμων δεν θα πρέπει να είναι πρόσχημα για να αγκαλιάσουμε τις ε, τεχνολογίες γενετικών τροποποιημένων τροφίμων. Διότι εν δυνάμει θα μπορούσε να είναι πολύ επικίνδυνα. Υπάρχουν πολλές ε, μελέτες άλλωστε που δείχνουν ότι οι πολίτες μας ε, δεν ζητούν γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Η εξάρτηση από τη βιοτεχνολογία άλλωστε μειώνει τη βιοπικιλότητα και μπορεί να οδηγήσει σε α, μεγαλύτερη αύξηση των ασθενειών και συγκέντρωση ε, ευρεσιτεχνιών στα χέρια μεγάλων ε, βιομηχανιών. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την δημιουργία νέων γενετικά τροποποιημένων ε, φυτών και τροφίμων, ε, διότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει απαράδεκτους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Άλλωστε η μείωση των πόρων ε, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην ε, κατάχρηση ή στην κακή χρήση της βιοοικονομίας. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέω κουσέ. Εδώ και ορισμένες εβδομάδες είχαμε την ανακοίνωση της Επιτροπής ε, και γίνεται λόγος για βελτιστοποίηση της χρήσης και της μεταχείρισης των αποβλήτων, να αποφύγουμε ε, τα αέρια θερμοκηπίου, αλλά μιλάμε για sustainable, για βιώσιμο για προϊόντα bio, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι μετά το Ρίο ε, το, το 92 έγινε μεγάλη πρόοδος στον κόσμο. Και αυτό αφορά και την ανακοίνωση και την έκθεση. Γίνεται ε, μία ρητορική εξισορρόπηση και προσπαθούμε να φιλοτεχνίσουμε κατά πράσινο τρόπο τα πάντα. Δεν μιλάμε για την αρχή της προφύλαξης, δεν γίνεται καμία ε, ε, επίκριση στα βιοκαύσιμα, γιατί ξέρουμε ότι και από πλευράς περιβάλλοντος και ενέργειας αποτελούν κάκιστο προηγούμενο και δεν μιλάμε για τους κινδύνους των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών ή τους κινδύνους της ε, νανοτεχνολογίας. Πρόκειται για μία ε, ε, ένα χρυσιθυρικό όραμα και μιλάμε για οικονομία bio κάτι το οποίο υποτίθεται ότι είναι πανάκια για όλα. Ακολουθεί η Κομισιόν. Η Αμπάλτσι. Είναι εδώ. Έχετε να προσθέσετε. Επικεφαλής της Μονάδας Βιοτεχνολογίας στη Σχετική Γενική Διεύθυνση. Έχετε το λόγο. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο Κοινοβούλιο για την βιοοικονομία και εκτιμά την έκθεση του εισηγητή. Ιδιαίτερα συμμεριζόμαστε το όραμα της Επιτροπής σας για τη μετάβαση προς μία βιώσιμη βιοοικονομία για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και για να συνεισφέρουμε στη δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομικής βιώσιμης ανάπτυξης. Η στρατηγική για τη βιοοικονομία βασίζεται στη χρήση ε, βιολογικών πόρων που να είναι πιο καινοτόμα και βιώσιμη, βιώσιμη από πλευράς περιβάλλοντος και οικονομίας. Μιλάμε για παραγωγικά συστήματα που να βασίζονται σε εξισορροπημένα και ανθεκτικά οικοσυστήματα. Να βασιζόμαστε στην χρήση ανανεώσιμων όπως ε, βιοδιηληστήρια και ανάπτυξη της, ε, και πρόθεση της απασχόλησης. Πρόκειται για καινοτόμα στοιχεία που είναι ύψης της σημασίας και ε, ευχαριστούμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για την ε, υλοποίηση αυτής της στρατηγικής λαμβάνοντας υπόψη και τις καινοτομίες. Τονίζουμε την αναγκαιότητα ενίσχυσης και προώθησης συνεργειών στους προσήκοντες τομείς της οικονομίας, οικονομίας πολιτικής συνοχής ΚΑΠ ορίζοντας 2020. Θα πρέπει να καταβληθούν κοινέ προσπάθειες όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά σε περιφερειακό και τοπικό. Μιλάμε για έρευνα και καινοτομία αλλά θα πρέπει να αναπτύξουμε και νέες αρμοδιότητες και γνώσεις μέσω ε, πολυεπιστημονικών σχέδιων κατάρτισης. Οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν επικαιροποιημένες ε, πληροφορίες για τη βιώσιμη κατανάλωση και να γίνονται γενικότερες συζητήσεις για τη βιοοικονομία. Τονίζουμε τη στρατηγική σημασία προώθησης πληροφοριών για τα νέα βιολογικά προϊόντα. Όπως ε, τονίζει και η Επιτροπή σας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, μεταφορά γνώσεων, κάτι το οποίο αφορά και τη σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Αυτή η εταιρική οικονομική σχέση θα προωθήσει νέες αλυσίδες αξιών με βάση βιολογικά προϊόντα. Τέλος, θα ήθελα να σας τονίσω ότι η Επιτροπή έχει προωθήσει ένα παρατηρητήριο για την βιοοικονομία στην Ευρώπη και προωθεί και ένα σχετικό πάνελ. Θα θέλαμε να παρακολουθήσετε τις ε, διεργασίες αυτές του παρατηρητηρίου και του πάνελ. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για μια βιώσιμη ε, βιοοικονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Μπαλτσί. Ο εισηγητής λαμβάνει πάλι το λόγο για να προβεί σε σύνοψη και να απαντήσει ενδεχομένως σε ερωτήσεις. Κύριε Μπαρτολότσι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που παρενέβησαν, ιδιαίτερα τους σκιώδεις και τις συνεισφορές όλων καθώς και τα σχόλια. Μερικά τα συμμερίζομαι πλήρως, ιδιαίτερα τις προτάσεις της κυρίας Μέρκης, για να έχουμε ενιαία θηρίδα και να εισαγάγουμε νέες πολιτικές για τις ΜΜΕ που είναι ύψης της σημασίας για τις πολιτικές αυτές. συμμερίζομαι και ορισμένες παρατηρήσεις που υπογραμμίζουν τον επίγοντα χαρακτήρα, δηλαδή να δώσουμε κίνητρα για την βιοοικονομία. Και αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν στην πρόταση ψηφίσματος να ορίσω τον επίγοντα χαρακτήρα αυτής της πολιτικής. για να κινήσουμε και την ε, ευρωπαϊκή διαδικασία προώθησης των βιομηχανιών, να δώσουμε νέες ευκαιρίες στην ε, βιοοικονομία. Πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος μπορεί να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. Θεωρώ λοιπόν ότι όλες οι πρωτοβουλίες και οι υποδείξεις που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη. Και όλα αυτά τα συνδέουμε με την ανάγκη μιας ε, ανάπτυξης ε, κάπως διαφορετικής που να συμβαδίζει με το περιβάλλον και με την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Νομίζω ότι υπ' αυτή την έννοια μπορούμε να προβλέψουμε και προώθηση της απασχόλησης. Νομίζω ότι η Ευρώπη έχει κάπως καθυστερήσει. Θα πρέπει να δώσουμε μια νέα όθηση έτσι ώστε να προωθήσουμε πραγματικές πολιτικές, διότι μέχρι τώρα χρηματοδοτούσαμε την έρευνα, μελέτες για την βιοοικονομία. Τώρα όμως που υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μια σοβαρή προσπάθεια να περάσουμε στην επιχειρησιακή φάση ευαισθητοποίησης της αγοράς, υποστηρίζοντας πραγματικές πρωτοβουλίες παραγωγικών διαδικασιών που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό νομίζω ότι απλώς πρέπει να σας πω ότι είμαι στη διάθεσή σας ε, για περαιτέρω διευκρινήσεις αν τις ε, επιθυμείτε και ελπίζω και κατά την επόμενη φάση υποβολής των τροπολογιών θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να θέσουμε σε εφαρμογή αυτή την θετική προσέγγιση μέσα στα πλαίσια της συζήτησης αυτού το μέλλον. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε τις τελικές αυτές παρατηρήσεις. Μιλήσατε και για τροπολογίες. Η προθεσμία κατάθεση είναι 27η Τρίτου. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα ψηφίσουμε στις 29 Μαΐου και ενδεικτικώς προβλέπεται η Ολομέλεια για την εκθεσή σας τον Ιούνιο. Ευχαριστώ όλες και όλους που αντέξατε μέχρι τέλους, που συζητήσατε το θέμα σας εύχομαι καλή ανάπαυση και θα τα πούμε αύριο στις 10 και οι συντονιστές μία ώρα πριν διακόπτουμε τη συνεδρίαση.